Sí. Buenos días a todos. Καλημέρα σε όλους. Σας παρακαλώ καθίστε. Είναι εδώ ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο κύριος Πίτερς, και θα ξεκινήσουμε με αυτό το σημείο της μερίσιας διάταξης, την παρουσίαση της ε, Βελγικής Προεδρίας. Ε, να καλωσορίσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Πέτερς. Όπως ξέρετε, είμαστε στην αρχή της Βελγικής Προεδρίας και ο κύριος Πέτρης βρίσκεται εδώ ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Εγώ έχω γνωρίσει τον κύριο Πέτερς από το άτυπο συμβούλιο του Βίγκο, στο οποίο συμμετείχα ως πρόεδρος της Επιτροπής μας και ο κύριος Πέτερς ε, διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το άτυπο συμβούλιο και όπως ε, γνωρίζετε η Βελγική Προεδρία συμπίπτει με ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας, τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής δηλαδή ε, όλες τις διαδικασίες συναπόφασης που έχουμε ξεκινήσει, οι οποίες καθυστέρησαν ε, και στη διάρκεια της ε, Ισπανικής Προεδρίας και ελπίζουμε να επιληθούν όλα αυτά τα θέματα στη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας. Θα ήθελα εξ ονόματος ε, της Επιτροπής μου να σας θέσω δύο θέματα, τα οποία ελπίζω να συζητήσετε στη διάρκεια της παρέμβασής σας. Και το ένα αφορά τη διαδικασία συναπόφασης και τα πολιετή σχέδια και το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με τη νομική βάση ε, που έχουμε για τα δύο σχέδια τα οποία είναι επιτάπτως αυτή τη στιγμή του Γαύρου και του Σαβριδιού ε, και το Συμβούλιο διαφωνεί με την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη θέση, διότι αυτοί οι αρμοδιότητες μας δίνονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το θέμα, εγώ εχθέ είπα ότι αυτό είναι Κάσιους μπέλι. Βέβαια δεν θέλω να είμαι τόσο σκληρή και να αναφέρομαι σε Κάσιους μπέλι, αλλά αν δεν επιληθεί θα ήθελα να σα επισημάνω ότι το θέμα αποτελεί προτεραιότητα για μα και είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε μέχρι τέλους. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο ίσως ε, να σα διαφεύγει, είναι το θέμα τη έντονη αντίθεση που έχει το Συμβούλιο και απευθύνομαι σε εσά ω Προεδρεύον του Συμβουλίου για να δούμε αν μπορείτε να κάνετε κάτι για το θέμα της συμμετοχής ε, των ευρωβουλευτών ε, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αλίας ως παρατηρητές όχι μόνο στις πολυμερείς συμφωνίες αλλά και στις διμερείς συμφωνίες. Υπάρχει μια σαφή θέση του Συμβουλίου, εμείς δεν κατανοούμε γιατί υπάρχει αυτή η θέση, δεν θέλουμε να είμαστε παρόντες στις διαπραγματεύσεις, θέλουμε απλώς να είμαστε παρατηρητές ε, όπως και το Συμβούλιο το οποίο δεν διαπραγματεύεται επίσης και δεν καταλαβαίνουμε γιατί έχει τόσο αυστηρή στάση το Συμβούλιο και γιατί το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είναι πολύ αρνητική και η δική μα εστιάση σε ε, συμφωνία αυτή πλαίσιο. Θα συνεχίσουμε να ε, κυνηγάμε αυτό το θέμα και ε, ελπίζω να μπορέσετε να διαδραματίσετε κι εσείς κάποιο ρόλο ώστε να είναι λίγο πιο ευέλικτη η θέση του Συμβουλίου επί του θέματος. Μετά από όλα αυτά να σας καλωσορίσω, να σας δώσω το λόγο και κατόπιν θα δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους ευρωβουλευτές που θέλουν να σας θέσουν ερωτήσεις να παρέμβουν. Σας ευχαριστώ λοιπόν, καλωσορίσατε και έχετε το λόγο. mevrouw de voorzitter. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να εκπροσωπήσω την ε, ε, επερχόμενη Προεδρία για τους επόμενους έξι μήνες δηλαδή και θέλω καταρχήν να σας πω πόσο ενδιαφέρομαι και επίσης ε, η ε, βελγική κυβέρνηση για τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην νομοθετική διαδικασία στον τομέα της αλληλείας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχω ήδη συζητήσει με την Πρόεδρό σας και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να υπενθυμίσω πόσο θεωρώ ότι είναι βασικός ο, ο ρόλος της Επιτροπής σας. Τώρα που συνεργαζόμαστε στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, θα ήθελα επίσης να συγκεκριμενοποιήσω τη συνεργασία μεταξύ μας κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν γρήγορα οι τα διάφορα θέματα τα οποία είναι η προσυζήτηση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την απερχόμενη Προεδρία κυρία Εσπινόζα για την εξαιρετική εργασία της, διότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της πολλά θέματα καλύφθηκαν και κατέληξαν και πιστεύω ότι συμφωνήσατε μαζί της σε ένα πλαίσιο που αναφέρεται στην τακτική νομοθετική διαδικασία. Άλλωστε, ε, διήφθηνε το Συμβούλιο για την ε, αναθεώρηση της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής και της οργανώσεως της κοινή αγοράς. Θέλω να την ευχαριστήσω για όλα αυτά. Όπως ξέρετε υπάρχουν διάφορα σημαντικά θέματα της αλληλείας τα οποία θα ήθελα να συζητηθούν στα Συμβούλια του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Μεταξύ των προτεραιοτήτων αναφέρομαι εις τις ε, ποσοστώσεις και, και τα τάκ για το 2011 στην αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και στην πρόοδο των πολιετών διαχειριστικών προγραμμάτων. Είναι δηλαδή ένα μείγμα από βραχυπρόθεσμες, μακρυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δραστηριότητε. Επειδή αναφερόμαστε εις τις δυνατότητες αλίας για το 2011, ήθιστε για κάθε προεδρία ε, του δευτέρου εξαμήνου του έτους να αντιμετωπίζει το γεγονός ότι σύντομα θα πρέπει να καθοριστούν τα επίπεδα των αλλιευμάτων για το επόμενο έτος και εφόσον εδώ μιλάμε για τα ΤΑΚ και τις ποσοστώσεις για το 2011 θα βασιστώ σε ορισμένες αρχές τις οποίες θέλω να παρουσιάσω τώρα. Καταρχήν, θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός προσοδοφόρου τομέα. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο διότι όσο έχει κατάσταση τώρα, ε, δηλαδή με την οικονομική κρίση, τα εισοδήματα των αλλιέων ε, κινδυνεύουν και πιέζονται. Συγχρόνως όμως πρέπει να υπάρχει μία υφόρα εκμετάλλευση των αλλιευτικών αποθεμάτων και διότι εξαρτάται από αυτά η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κατάσταση του εισοδήματος των αλλιέων και θα πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο τομέων και όσο και να έχουμε πείρα δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή. Δεύτερον, ε, η ιδέα μας είναι ότι τα ΤΑΚ πρέπει να βασιστούν σε ε, μία επιστημονική ε, γνωμοδότηση, πράγμα όμως το οποίο ε, δεν είναι ίσως προφανές. Και υπάρχει ένα θετικό στοιχείο. Τα επίπεδα που καθορίσαμε πέρυσι ε, προσέγγιζαν περισσότερο την επιστημονική γνωμοδότηση από ό,τι στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, οι πόροι για τους οποίους δεν έχουμε ε, επιστημονική γνωμοδότηση αυξάνονται και παρόλο που επενδύουμε πολλά χρήματα και το 2008 καταρτήσαμε ένα νέο πλαίσιο συγκεντρώσεως των στοιχείων. Θα επανέλθω όμως στα θέματα αυτά. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ εις ε, τα μακροπρόθεσμα διαχειριστικά προγράμματα τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί διότι πρόκειται ε, ε, για θέματα τα οποία υφίστανται συχνά βραχυπρόθεσμη πολιτική πίεση για να αποκλίνουμε από αυτά. Οπότε αυτό πρέπει να σταματήσει. Όπως ξέρετε θέλουμε να συνεργαστούμε την Επιτροπή για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Ορβηγία πριν από το τέλος του 2010. Διότι ήδη πέρυσι είδαμε πόσο δυσάρεστη μπορεί να είναι η κατάσταση εάν δεν έχουμε συμφωνήσει με την Ορβηγία μέχρι το τέλος του έτους. Και γι' αυτό κυρίες και κύριοι συνοψίζω ότι αποβλέπουμε σε μία πολιτική συμφωνία με τα, ε, για τα τάκα της Βαλτικής για το 2011 στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου, για τα τάκα της Ανοιχτής Θαλάσσης ε, για το 2011 και 2012 στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου και τα βασικά τάκ και της ποσοστός για το 2011 καθώς και τα τάκ της Μαύρης Θάλασσας για το 2011 στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Δεύτερο βασικό θέμα για την ε, Βελγική Προεδρία είναι η αναθεώρηση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής διότι η Προεδρία μας δεν προβλέπει να λάβει τυπικά μέτρα για να, αναθεωρήσει την κοινή αλληλευτική πολιτική. Αλλά σκοπεύουμε να διευκρινίσουμε τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διαδικασία αυτής. Γι' αυτό και θα οργανώσουμε ένα συμπόσιο το οποίο ε, θα ασχοληθεί με μία από τις βασικές ε, σχέσεις ε, στον τομέα της αλληλείας, δηλαδή μεταξύ αλληλείας και επιστημόνων μπορούμε να βελτιώσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο εμπλεκομένων για να μπορέσει να προχωρέσει η αλληλευτική πολιτική και πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι ε, το θέμα της εργασίας των περιφερειακών συμβολίων. Πρέπει όμως να σας πω ότι ε, πολλές φορές ε, ε, δίστανται οι γνώμες μεταξύ επιστημόνων και ειδικών της αλληλείας όσον αφορά το μέλλον της αλληλείας και της διαχειρίσεως του περιβάλλοντος, πράγμα το οποίο τροφοδοτεί τη συζήτηση και γι' αυτό θα χρειαστεί ε, μία στρατηγική η οποία να συγκεράσει όλες τις πτυχές. Το συμπόσιο αυτό το οποίο έχει σαν τίτλο την αλληλεία, ε, βελτιωμένη αλληλεία και ε, συνεργασίες επιστημονικές για να οδηγήσουν την πολιτική. Θα οργανωθεί 9 και 10 Νοεμβρίου στην Οστάνδη για να συζητηθούν τα θέματα και να παρουσιαστούν τα πορίσματα στους Υπουργούς στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου όπου θα συζητηθούν, ελπίζω. Ελπίζω επιπλέον κυρία Πρόεδρε, ότι όπως και τα μέλη της Επιτροπής σας ε, ε, θα συμμετάσχετε σε αυτό το συνέδριο και θα μας τιμούσε ιδιαίτερος η παρουσία σας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα συναντηθούμε εκεί και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Επόμενο θέμα τα προγράμματα πολυ, ε, του προσανατολισμού και αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων που είναι ο τρίτος πυλώνας δραστηριότητος της Βελγικής Προεδρίας για τον τομέα της αλληλείας. Είναι βασικό να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ε, ε, για την, τον Γαύρο, και ε, το ε, το Σαφρίδι διότι για πρώτη φορά έχουμε ε, να ασχοληθούμε με ένα θέμα που βρίσκει την σύμφωνη γνώμη των επιστημόνων και της βιομηχανίας και μόνο έτσι θα μπορέσει να έχει ένα καλό μέλλον η αλληλεία ε, και να εξασφαλιστεί ο αηφόρος χαρακτήρας των πόρων. Επίσης θα πρέπει να καταμερίσουμε τις ε, αρμοδιότητες μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων αλλά πιστεύω ότι τα προβλήματα αυτά δεν είναι ανυπέρβλητα και θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Όσον αφορά το πολιετές πρόγραμμα για το Γαύρο δεν είναι λιγότερο σημαντικό από ότι αυτά που προανέφερα και αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι ένα πολιτικό πρόβλημα πολύ ευαίσθητο όπως απέδειξαν οι νυχτερινές συνεδριάσεις του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο αλλά για όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στον έλεγχο ελπίζω ότι θα παραμείνουμε στο πλαίσιο του κανονισμού ελέγχου πράγμα το οποίο θα διευκολύνει το έργο μας όσον αφορά τον έλεγχο των αλλιευμάτων όταν ε, ε, ε, φτάνουμε στο επίπεδο ασφαλείας θα πρέπει να αξιολογήσουμε το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου και να συγκεράσουμε τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη με την περιβαλλοντολογική αηφορία. Ξέρω ότι είναι βασικό να καθορίσουμε αυτό το ποσοστό και ε, θα προσπαθήσω να ε, φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Επίσης θα ήθελα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ε, ε, και κατά την Προεδρία μας και μετά θα ασχοληθούμε ε, με τα πολιετή προγράμματα για τον Σολομό στην Βαλτική. Και τέλος κυρία Πρόεδρε θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο το πολιετές πρόγραμμα για τα επίπεδα ψάρια στην Βόρειο Θάλασσα και ελπίζω ότι θα το επιτρέψουμε επιτύχουμε γιατί πρόκειται ε, για πολύ ε, βρασικά ε, θέματα και για τον δικό μας στόλο ένα άλλο βασικό θέμα είναι η εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, όπου για πρώτη φορά πρέπει να αξιολογήσουμε τα μεταβατικά μέτρα για την ρύθμιση των τάξ στη Βαλτική. Και για πρώτη φορά θα ισχύσουν ε, τα μέτρα αυτά στα πλαίσια της Βαλτικής. Για να μην υπάρξει ένα νομικό κενό. Θα πρέπει τα μέτρα αυτά να έχουν υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του χώρου, χρόνου και ε, ε, θέλω να ελπίζω ότι θα με στηρίξετε επικοδομητικά. Το δεύτερο θέμα είναι ε, η διαβούλευση για τεχνικά μέτρα στη Βόρειο Θάλασσα και τον Ατλαντικό, διότι θα εκπνεύσουν του χρόνου τον Ιούνιο και είναι πολύ βασικό να προχωρήσουμε σε αυτό τον φάκελο κατά τρόπον ώστε όταν οι Ούγγροι ε, θα ολοκληρώσουν ε, αυτό το θέμα να μπορέσουν ε, να καταλήξουν σύντομα. Τέλος, το τελευταίο, τα τελευταία θέματα είναι τα εξωτερικά. Έτσι θα τα χαρακτήριζα. Διότι όπως ξέρετε όταν το φθινόπωρο πρέπει να διαπραγματευτούμε βασικά θέματα για την αλληλεία το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι πολύ βεβαρημένο. Ήδη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα ετοιμάσουμε τις ετήσιες διαπραγματεύσεις με την Νορβηγία. Η ΕΚΑΤ έχει επίσης μεγάλη σημασία ε, γιατί θα πρέπει να δοθεί εντολή στο Συμβούλιο για την διαπραγμάτευση για τον ερυθρό τόνο την ετήσια συνάντηση στο Παρίσι. Ξέρουμε ότι οι προετοιμασίες για το Παρίσι θα είναι δύσκολες διότι θα χρειαστεί να τέμνουμε γόρδιους δεσμούς και γι' αυτό θα προωθήσω μια καλή συνεργασία μεταξύ αλλιέων και επιστημόνων. Και τέλος θα έχουμε την πρόκληση της ε, αρχής των διαπραγματεύσεων της Ισλανδίας για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη και αν δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητός μας η αλληλεία θα είναι ένα βασικό και ίσως κεφαλαιόδες θέμα για την διαδικασία αυτή προσχωρήσεως άρα θα ακολουθήσουμε ε, εκ του σε αυτό το θέμα. Κυρίες και κύριοι, ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι βλέπετε ότι το πρόγραμμά μας είναι πάρα πολύ ε, βαρύ ε, για το δεύτερο εξάμεινο και ξεκινάω από την αρχή ότι μετά από ένα ωραίο καλοκαίρι όλοι θα είμαστε φρέσκοι και ενθουσιώδεις για να μπορέσουμε να αφιερωθούμε στην εργασία μας διότι ο άμεσος χρόνος θα είναι πολύ βασικός για να υπάρξει μία η ανάπτυξη και συνεργασία. Ένα-ένα τα προγράμματα θα μπορέσουμε να τα προωθήσουμε για να καταρτήσουμε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διαχειρίσεως που θα εξασφαλίσει ένα σωστό εισόδημα στους αλληλείς μας και ευρωπαϊκό ψάρι για τα παιδιά μας. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμη η Προεδρία μας, οπότε σας ευχαριστώ ε, για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους ε, συντονιστές, όσους ε, ήθιστε. Θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο συντονιστών. Αν θέλετε, στις μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπου ε, βουλευτές που θα ζητήσουν το λόγο και αν θέλετε να φύγετε θα με ενημερώσετε και θα επιταχύνουμε τα πράγματα. Καταρχήν η κυρία Πετράκ, μέρος του ΕΛΚ. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω καλημερίζοντας τον κύριο Υπουργό και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για τα καθήκοντά σας στο πλαίσιο της Βελγικής Προεδρίας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας στο σύνολό της. Μας παρουσιάσετε εδώ μια γεμάτη ατζέντα, αλλά ρεαλιστική θα έλεγα πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε πολλές φορές να παρουσιαστούν πάρα πολύ φιλόδοξα σχέδια και βλέπουμε ήδη από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελοπιθούν. Στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι παρόλο που είναι γεμάτη η ατζέντα σας είναι ρεαλιστική και λογικά θα μπορέσετε να την υλοποιήσετε. Είναι ένα σημείο αρκετά θετικό. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής σας ανοίγεται ε, μια θεματική εγκάρσια και είχε να κάνει με, μεταξύ, με τη σχέση μεταξύ ε, αλλιών και επιστημόνων και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Αυτό ήταν ε, παρόν σε όλη σας την παρέμβαση. Μπορώ να σας πω ότι αυτό αποτελεί ανησυχία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα η έκθεση για την ε, πράσινη βίβλο, για την μελλοντική μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΛΠ. Θεωρούμε ότι έχουμε τρεις πυλώνες που είναι και ο περιβαλλοντικός, ο οικονομικός και ο κοινωνικός και πρέπει να του διατηρήσουμε. Έτσι λοιπόν σε όλες τι θεματικές που θα προσεγγίσετε αυτό θέλουμε να διατηρηθεί. Είπατε είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Αναμφισβήτητα όμως αυτή η δύσκολη οδό είναι αυτή που θα παρέσει να μα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Και έτσι λοιπόν αυτή την οδό πρέπει να ακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν θα ήθελα τώρα να τονίσω αυτό που αναφέρθηκε ως προοπτικές ε, των αλλιέων και των επιστημόνων. Πολλές φορές οι απόψεις ε, των δύο ε, δεν συναντώνται. Έτσι λοιπόν εδώ είναι, έχουμε και ένα θέμα επικοινωνίας. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο και αν ασχοληθεί η Βελγική Προεδρία με το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι δυνατόν να βελτιώστε την επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων και ελαίων και την εγκύτητά τους, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για την ε, αηφορία της αλίας και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσετε αυτές τις ε, μορφές επικοινωνίας μεταξύ τους. Αναγνωρίζουν οι αλίες ότι πρέπει να ε, υπάρχει ουσιαστικά βιωσιμότητα στον τομέα της αλίας για το μέλλον. Και μία τελευταία πτυχή που ήθελα να αναφέρω εδώ έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ των τριών ε, οργάνων. Και εδώ πολύ συγκεκριμένα μιλάμε για τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν της θέσης ισχύ της συνθήκης Ελισαβόνα. Της Ελισαβόνας, με Φυσικά είναι πολύ σημαντικό από την αρχή καθώς τώρα θα μπούμε στο δεύτερο εξάμεινο που θα ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν από την αρχή οι σχέσεις μεταξύ των τριών οργάνων και ιδιαίτερα οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναγνωριστούν σαφώς από τους διάφορους οργανισμούς έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν, ε, να υλοποιηθούν πλήρως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, προέρχεται από άμεση ψηφοφορία, έτσι λοιπόν εκπροσωπεί περισσότερο τους πολίτες από τα υπόλοιπα όργανα και θέλουμε εμείς ε, να θέσουμε τις γενικές γραμμές ενδιαφέροντος για τον τομέα της Ελίας και θεωρούμε ότι η δική μας παρουσία σε όλους τους τομείς της Ελίας είναι πάρα πολύ σημαντική για το βιώσιμο μέλλον του τομέα. Έτσι λοιπόν μπορώ να σας πω ότι θα έχετε την πλήρη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά και εμείς θέλουμε και βασιζόμαστε στη δική σας επιρροή ε, για να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στα διάφορα φόρα έτσι ώστε οι συμφωνίες τις οποίες θα καταλήξουμε να έχουν ε, στο μέλλον αποτελεσματικό αντίκτυπο. Αυτό έχει να κάνει με όλα τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε εδώ συγκεκριμένα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια βιωσιμότητας και επίσης για τις συμφωνίες με την Νορβηγία και την Ισλανδία. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, στις 14 πρέπει να φύγει ο κύριος Υπουργός. Ναι κύριε Ρόντους, τώρα θα σας δώσω το λόγο. Απλώς θέλω να σας πω, παρακαλώ, σεβαστείτε τον χρόνο των τριών λεπτών για τους συντονιστές και θα δούμε πόσο χρόνο θα έχουμε και για τα υπόλοιπα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Ρόντουστ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ κύριε Υπουργέ θέλω να σας καλωσορίσω και χαίρομαι για αυτά που μόλις είπατε. Θα είμαι πολύ σύντομη και θα παρουσιάσω ε, πολύ συνοπτικά τις παρατηρήσεις ε, μου. Χαίρομαι που συνεργάζεστε έντονα με ε, την επιστήμη διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ελέγξουμε την αλληλεία. Χαίρομαι που έχετε αυτή την πρόθεση αλλά πιστεύω ότι πήρα των ε, αλλιέων πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και να βρεθούν τρόποι κατά τρόπον ε, ώστε ε, να μπορεί να τα καταφέρει και ο αλλιέας, δηλαδή να σεβαστεί τα στοιχεία αυτά. Θα ήθελα να έχετε τα στοιχεία των αλλιέων, αλλά αντιλαμβάνουμε ότι αυτή είναι επιφυλακτική και ίσως εκεί θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί πείτε πράγμα για το οποίο θα σας είμαι ευγνώμων εάν το πράξετε. Όσον αφορά το συμπόσιο, θα ευχαρίστω θα δεχθώ την ε, πρόσκλησή σας και ελπίζω ότι θα έρθουν και οι συνάδελφοι για να συζητήσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα. Καταρχήν τη διαδικασία προσχωρήσεων της Ισλανδίας, όπου σαν Επιτροπή Αλληλείας θα πρέπει ακόμη να λύσουμε διάφορα δύσκολα προβλήματα και προσβλέπω στη στήριξη γιατί η απέτηση των Ισλανδών να προστατεύσουν την αλληλεία τους και να μπορέσουν να προχωρήσουν στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα διαπραγματευτούμε και ελπίζω ότι συσπηρωμένοι ε, θα επιτύχουμε κάτι παραπάνω από ό,τι αν αποκλείει ο ένας τον άλλον. Και όσον αφορά την αμοιβαία, τον αποκλεισμό. Ήθελα να σας πω ότι ε, περιγράψατε για μας ότι η, ε, ε, κάτι που είναι μεγάλο πρόβλημα για αυτή την Επιτροπή και παραπέμπω εδώ εις την κατάληξη της κυρίας Φράγκα προηγουμένως. Δηλαδή είμαστε πολύ θυμωμένοι διότι το Συμβούλιο δεν έχει δεχθεί να συμμετέχουμε σαν παρατηρητής στις διαπραγματεύσεις, πράγμα το οποίων δικαιούμαστε σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και χθε συζητήσαμε ε, ε, ενδελεχώς το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν θα δεχθούμε. Δεν μπορείτε να μας αποκλείετε και θέλω στο σημείο αυτό επίσης να σας πω ότι οι συμφωνίες αλληλείας αποτελούν πάντοτε ένα πρόβλημα στην Επιτροπή ε, αυτή διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, την περιβαλλοντολογική αηφορία, τα οικονομικά συμφέροντα και θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι για να καταλήξουμε σε σωστές αποφάσεις και σε όλα αυτά σας εύχομαι καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε κύριο Γκάλαγκερ για τους φιλελευθέρους, ο οποίος είναι και εισηγητής για το πολιετές ε, σχέδιο για το Σαφρίδι. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσω τον κύριο Υπουργό και να τον ευχαριστήσω που μας παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας ε, για τους επόμενους έξι μήνες. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας. Ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, έτσι λοιπόν ε, δεν θα αναφερθώ σε πολλά από αυτά που αναφερθήκατε για τα τακέτες ποσοστώσεις, ε, για την θεωρήση της κοινωνιστικής πολιτικής. Δεν θεωρώ ότι θα συνεισφέρετε ε, πάρα πολύ σε αυτό, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένα θέματα για τα οποία εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τον κλάδο κατά τους επόμενους μήνες. Είμαστε σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση αυτή τη στιγμή ε, σε σχέση Norway, με το σκουμπρί. Ε, ξέρετε ότι αλλιεύεται αυτό και στην Ορβηγία και από την Ισλανδία. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε το πόθεμα, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι βιώσιμο όλο αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας και αναφέρθηκα στις δυσκολίες που προέκυψαν πέρσι το Δεκεμβρίο με την Ορβηγία αλλά ε, από ό,τι κατάλαβα τώρα αυτό το θέμα έχει επιληθεί για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχουμε ε, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το θέμα αυτό γιατί αύξησε η Ισλανδία την ποσόστοση από 4.000 σε 130.000 τόνους, ε, δηλαδή έχουμε αύξηση επί 40 και μιλάμε για το ίδιο απόθεμα επί το οποίο εξαρτώμαστε και εμείς. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Συμφωνία Προσχώρησης, γιατί αν η Συμφωνία Προσχώρησης ε, χρειαστεί ε, διαρκήσει για 10 χρόνια, τότε δεν θα υπάρχει σκουμπρί σε 10 χρόνια και αυτή είναι μια μονομερής απόφαση που ελήφθη από την Ισλανδία και εγώ πιστεύω ότι πρόεδρε έχετε εδώ ένα ρόλο να διαρματίσετε και να συνεργαστείτε με την Δαμανάκη, η οποία έχει λάβει κάθε τη θέση και από ό,τι κατάλαβα ε, ήθελε να θέσει ως όρο για τις συνομιλίες ε, προσχώρησης να έχει επιληθεί το ζήτημα αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι η Προεδρία σας θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και θα ήθελα εσείς να εμπλακείτε τα μάλα. Σε ό,τι αφορά τώρα το σκουμπί στο οποίο αναφερθήκε η Πρόεδρος, ε, εγώ συναντήθηκα με το Συμβούλιο, πραγματικά συνεργαστήκαμε και μπορώ να σας πω ότι ε, αν δεν θα είχαμε πρόβλημα ε, ευτυχώς Προβλανδοί δηλαδή ψήφισαν ναι στη συνδίκη Αβώνας αλλά τώρα ε, μπορώ να σας πω ότι έχουμε καταλήξει σε μια προβληματική κατάσταση. Εμείς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τις συμβουλώσεις. Σχεδόν τα έχουμε καταφέρει, αλλά τώρα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση ότι η συμβουλή, η γνωμοδότηση που έλαβε το Συμβουλίο, πάνω από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να μην ήταν αυτό που θέλω να ακούσουν. Δηλαδή τώρα όμως το Συμβούλιο δεν μπορεί να έχει και την πίτα ολόκληρη και τη σκυλοχορτάτο ήταν ε, το θέμα της νομικής βάσης η 43.2. Εμείς ε, κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να ε, έχουμε ρόλο για τα τάκια της ποσοστώσης, αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να το επιλύσουμε αυτό. Και να σας πω, όταν δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στην επιστήμη, τόσο σημαντικές είναι και οι πληροφορίες που μπορούν να δώσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, στους επιστήμονες. Εγώ νομίζω ότι συνεργάζονται και στο παρελθόν ε, έχουμε δει ότι ε, τα συστήθηκαν τα ΡΑΚ, τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβουλία, τα οποία είναι πάρα πολύ υπεύθυνοι φορείς και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, Πρόεδρε, εγώ αναμένω από εσά να βοηθήσετε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει να κάνει για το θέμα του σκουμπρού με την Ισλανδία. Ε, δεν θα αναφερθώ στο θέμα των ε, απορρίψεων. Ε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνει η δική σας Προεδρία, να ασχοληθεί δηλαδή με το θέμα αυτό και η επόμενη Προεδρία, για να το επιλύσουμε το συντομότερο. Τώρα, το να μιλάμε για μηδέν απορρίψεις ε, θα ήταν εντελώς μη ρεαλιστικό. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κάποια πρόοδο και να βοηθήσουμε και τους αλείς. Ευχαριστώ για τους πρασίνους η κυρία Λομπίν για τρία λεπτά. Tack så hemskt mycket och välkommen hit, eh, inkommande president. Det var väldigt intressant att höra. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσε ήταν οι προτεραιότητε που μα παρουσιάσατε για του επόμενου 6 μήνε. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΛ, από ό,τι φαίνεται παρουσιάζεται ως πολύ σημαντικό στοιχείο τη επιστημονικές ε, συμβουλές. Επίσης αναφέρεται ότι οι διαπραγματεύσεις για τα τάρκη της ποτοσυστώση και τα πολιετή προγράμματα θα ε, πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικέ συμβουλέ. Ε, το κάνατε να ακούγονται πάρα πολύ απλά, αλλά στην πράξη δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι εντοπίσατε τα κυρία προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω αυτό οδήγησε στην καταστροφική κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε πάνω από το 80% των αποθεμάτων ε, να την χάνουν εντατική εκμετάλλευση, υπερβολική εκμετάλλευση. Και αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι εκτό του ασφαλούς βιολογικού ορίου. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτές υποστημονικέ συμβολέ. συμβολές. Αναρωτιέμαι τι σκοπεύει να κάνει η Βελγική Προεδρία για να βελτιώσει την κατάσταση. Μια άλλη ερώτηση είναι εξή. Πώς η Βελγική Προεδρία πρόκειται να εργαστεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τα επόμενα τακτή ποσοστώσεις. Πώς θα ακολουθήσει τις επιστημονικές συμβουλές. Ξέρουμε ποιες είναι οι επιστημονικές συμβουλές. Φανταστείτε σε ποια κατάσταση θα ήμασταν τώρα αν ακολουθήσαμε τι επιστημονικέ συμβουλέ πριν 10 χρόνια. Νομίζω ότι θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα γιατί θα είχαμε και πολύ περισσότερα αποθέματα. Νομίζω ότι και ο λευτικό τομέα θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση σήμερα. Δεν Νομίζω ότι από την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα κερδίζει κανεί. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να μα πείτε κάποιε περισσότερε πληροφορίε για την ε, βασική στάση που θα ακολουθήσει η Προεδρία στο θέμα αυτό. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίξουμε τον κλάδο οικονομικά, αλλά θα ήθελα να τοποθετηθείτε για την υλοποίηση συμβασμών μεταξύ των κλάδων. Πώς ε, ουσιαστικά θα συνδέασετε τα βραχυπρόθεσμα αιτήματα με το μακροπρόθεσμο θέμα της ε, βιωσιμότητας του τομέα. Και κάτι που δεν, δεν άκουσα μάλλον από την παρουσίασή σας ήταν για το πόσο κακή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη τώρα. Στην Ευρώπη έχουμε θάλασσες όπου γίνεται η μεγαλύτερη περιελήψη στον κόσμο. Εσείς ε, αναλαμβάνετε την Προεδρία στα μέσα της μεταρρύθμισης και νησιλευτικής πολιτικής και θα πρέπει να ασχοληθείτε με τα θέματα αυτά. Ο κ. Γκάλακερ έκανε ένα πολύ καλό σχόλιο για τις απορρίψεις αναφερθήκατε και εσείς αυτό. Θα πρέπει να απορρίψουμε την ιδέα ότι μπορούμε να απαγορεύσουμε πλήρως τι απορρίψει. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέλαμε να είναι παρατηρητή σε όλες τις διμερεί ε, διαπραγματεύσει. Ε, ευχαριστώ.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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας. Ε, κύριε Υπουργέ, θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπατε και που θεώρησα πολύ βασικό, την έλλειψη επιστημονική πραγματικής ενημέρωση, Διότι πολλές φορές δεν έχουμε επαρκή στοιχεία και αυτό είναι κατανοητό. Βάσει λοιπόν αυτής της ελλείψεω ενημέρωση, πρέπει να λαμβάνονται πολύ σημαντικέ αποφάσεις που έχουν σχέση με ε, τις ποσοστώσεις, πράγμα το οποίο οδηγεί σε ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την αλληλεία και με το λογιστικό σύστημα και με το σύστημα ενημέρωσης ε, όταν προσπαθούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος των αποθεμάτων και αυτό χρειάζεται επιστημονική έρευνα. Οπότε από την άποψη αυτή προβλέπετε ότι θα οργανώσετε ε, στο συμπόσιο που θα οργανωθεί σαν ε, ε, προσπάθεια να καταρτίσετε μία αναθεώρηση της ε, κοινής αλληλευτική πολιτική, ότι αυτό θα είναι δηλαδή ένας από τους στόχους σα, διότι πρέπει να σας πω τι ανησυχίες μου νόμιζα ότι το πρόγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί και τώρα θα έπρεπε να δράσετε ε, διότι η έλλειψη δράσης ε, είναι ει βάρο των ε, αλλιέων και είναι προφανές ότι η αλληλευτική πολιτική δεν εφαρμόζεται σωστά. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι όταν μιλάμε για την κοινή αλληλευτική πολιτική βασιζόμαστε στη μεταφορά των ποσοστώσεων πράγμα το οποίο οδηγεί σε εκνευρισμούς ανησυχίες και περιπλοκές. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η θέση σας στο θέμα αυτό, δηλαδή πώς πρόκειται να το εφαρμόσετε αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις και σχόλιο και κατόπιν θα περάσουμε στον γύρο των υπολείπων ευρωβουλευτών πέραν των συντονιστών που μόλις ακούσαμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω όλους εσάς ε, για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ρεαλιστές και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με τον κατάλληλο τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς ε, αυτά που είπε η κυρία Πατράου είναι πάρα πολύ σημαντικά χρειάζεται να έχουμε τον κατάλληλο χρόνο στη διάθεσή μας, να εντοπίσουμε ποια είναι τα προβλήματα και από εκεί και πέρα να διαπιστώσουμε τι μπορούμε να προχωρήσουμε και τι μπορούμε να επιλύσουμε στο επόμενο εξάμεινο. Θα πρέπει βέβαια να γίνεται μια καλή ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας. Και με χαροποιεί το γεγονός ότι όλα όσα είπατε για το συμπόσιο και τις σχέσεις μεταξύ επιστημόνων και αλληλευτικού τομέα ε, φαίνεται να αρέσουν στην Επιτροπή σας και χαίρομαι που είναι κοινό το όραμα. Πολύ λογικά αναφερθήκατε και στα προβλήματα επικοινωνίας. Στο συμπόσιο θα υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία θα επισημανθούν και η επικοινωνία είναι ένα από τα θέματα τα οποία ε, θα συζητήσουμε και θα σταθούμε παραπάνω. Πολύ σωστά λοιπόν το επισημαίνετε ως ε, μία από τις βασικές μας ανησυχίες. Ετέθη επίσης μία ερώτηση από πλευράς κυρίας Ρόντους, η οποία πολύ σωστά μας είπε ότι Εάν ε, πρέπει να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων, τότε θα πρέπει να υπάρχει και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των αλλιέων. Αναφερθήκατε στα ημερολόγια σκάφους. Ε, νομίζω ότι στο συμπόσιο έχουμε την κατάλληλη ευκαιρία να γίνει ακριβώς αυτή η, ε, αυτό το άνοιγμα. Οι επιστήμονες και οι αλληλείς δεν συζητούν μεταξύ τους, αλλά αν τους συγκεντρώσουμε κάπου μαζί υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία θα μπορούσαν ίσως να καλύψουν. αναφερθήκατε σε κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη μιας τέτοιας συζήτησης. Κύριε Λεβίν, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι οι συζητήσεις για τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και οι ίδιες οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ε, είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι τόσο εύκολο να τις έχουμε. Υπάρχουν ανησυχίες για τα αλληλευτικά αποθέματα, ε, για τις ε, βιώσιμες δυνατότητες αλίας, αλλά ακριβώς εδώ διαδραματίζει ε, ουσιαστικό ρόλο η επιστημονική γνωμοδότηση. Και αυτή είναι συνεχή ανησυχία και στη διάρκεια τη Βελγική Προεδρία θα το συζητήσουμε, το να έχουμε κατάλληλε επιστημονικέ γνωμοδοτήσει, γιατί για κάποια αποθέματα αυτό είναι το ουσιώδες, να έχουμε τι κατάλληλε επιστημονικέ γνωμοδοτήσει. Πρέπει λοιπόν να το παρακολουθούμε και να το ενθαρρύνουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί εμεί είμαστε πεπισμένοι ότι η επιστημονική οδό είναι η μόνη οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε προκειμένου να επιτύχουμε βιώσιμη αλληλεία με αποτελεσματικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν ε, το θεωρούμε ικανή και αναγκαία συνθήκη και με χαροποιεί το γεγονός ότι συμφωνείτε και εσείς με αυτή την άποψη και υποστηρίζετε αυτή την άγουσα. Ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα το υλοποιήσουμε, στο συμπόσιο, το σκεπτικό μας είναι να κάνουμε μια αντιπαράθεση των επιστημονικών ονομαδοτήσεων με την πραγματικότητα που έχουμε από τον αλληλευτικό τομέα. Και θεωρώ ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να έχουμε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην πραγματικότητα ε, προκειμένου να επιτύχουμε τους συγκεκριμένου ε, στόχους που έχουμε στην πολιτική μας. Ο κύριος Γκάλεγκερ αναφέρθηκε στο σκουμπρί. Ναι, Πράγματι, μίλησα για το σκουμπρί στην πρώτη μου παρέμβαση. Ίσως θα μπορούσα να σας ε, εξηγήσω λίγο περισσότερο τα πράγματα. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε καταλήξει σε συμφωνία μέχρι το 2010. Νομίζω ότι αυτή ήταν η βασική σας ερώτηση ε, οι διαπραγματεύσεις με τα παράκτια κράτη, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία, τα νησιά Φαρόες και την Ισλανδία, ε, ήταν σε τέτοιο σημείο διεστάμενες που δεν φαινόταν να υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας μέχρι το 2010. Ε, η απέτηση της Ισλανδίας και των νησιών Φαρόες για πρόσβαση σε αλλιεύματα με πολύ ψηλότερο ποσοστό ε, δημιούργησε ε, έρηδες και φάνηκε να είναι... Ε, αντίθετη σε οποιαδήποτε παραχώρηση. Η Βελγική Προεδρία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τη προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία το φρινόπωρο, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο. Υποστηρίζουμε βέβαια παρόλα αυτά την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τα παράκτια κράτη να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Όπω και τα μέλη τη Επιτροπή σα, γνωρίζω πολύ καλά πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση για τα κρατημέλη που ενδιαφέρονται για αυτό το είδος και θα ήθελα να σας πω ότι η Επίτροπος στο Συμβούλιο της 20ης Ιουνιού δεσμεύτηκε να πιέσει την Ισλανδία και τα νησιά Φαρός και φυσικά θα τύχει της πλήρους υποστήριξής μου. και φυσικά η Προεδρία θα έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή και θα υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε, ενάντια σε χώρες που ε, κάνουν ανεύθυνη υπεραλίευση αυτών των αποθεμάτων. Αυτή είναι πάρα πολύ σαφής θέση και είναι η θέση της Προεδρίας μας. Τώρα λοιπόν, να περάσω στη σειρά των ερωτήσεων της μεταρρύθμισης κοινής ελευθερικής πολιτικής. Να πω εκ νέου ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2010 δεν θα έχουμε κάποια νομοθετική πρόταση που θα βασίζεται στην μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμεινο του 2011 που θα έχει αναλάβει τα Ινία η Ουγγρική Προεδρία. Όπως σας είπα λοιπόν, η δική μας συνεισφορά θα είναι το συμπόσιο το οποίο θα οργανωθεί και εδώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να κάνει και μια διάσκεψη για τη μεταρρύθμιση στις 16 Νοεμβρίου και η Βελγική Προεδρία θα ε, υποστηρίξει πλήρως ε, την εκδήλωση αυτή. Υπήρξε και κάποια ερώτηση για δράσεις. Όπως σας είπα, δεν υπάρχουν επίσημες προτάσεις ε, στο εξάμεινο της Βελγικής Προεδρίας. Εμείς βέβαια θέλουμε να καταλήξουμε σε μια απλή, εφικτή και πολύ στεναρή αλληλευτική πολιτική για το μέλλον. Έχουμε κάνει συζητήσεις επί του θέματος για τα οράματα και τις ευαισθησίες του καθενός εδώ και θα μπορούσα ίσως να σταθώ σε κάποιες από αυτές. Πέραν του γεγονότο ότι όπως σας είπα δεν θα έχουμε επίσημες προτάσεις, αυτές προβλέπονται για το πρώτο εξάμεινο του 2011. Η πολιτική για τα τάκια της ποσοστώσης θεωρούνται οι βασικές πολιτικές για την προστασία των αποθεμάτων, επομένως θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να τα διαχειριζόμαστε εύκολα να υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Υπάρχουν ε, κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την επιλεκτικότητα και το θέμα ε, των απορρίψεων. Η επικοινωνία μεταξύ αλλιών και επιστημονικού κλάδου θεωρείται βασική και επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ανανέωση του στόλου, τις χρηματοδοτήσεις και πώς μπορούμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό παραγωγικό τομέα. Θέλουμε να έχουμε μια ισχυρότερη οργάνωση αγοράς και να βοηθήσουμε τον αλληλευτικό τομέα κυρίως με τεχνικά μέτρα. Και επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, τον, ε, τις περιφερειακές ε, συμβουλευτικές οργανώσεις, τα ΡΑΚ. Επίσης αναφέρθηκε και το θέμα της μεταφοράς δικαιωμάτων, της ατομικής μεταφοράς δικαιωμάτων. Ε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει διάφορες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένες και της ε, εισαγωγής ενός τέτοιου συστήματος μεταφοράς ε, δικαιωμάτων. Κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Βίγκο, στο οποίο συμμετείχε και η πρόεδρο τη Επιτροπή σα, συζητήθηκε το θέμα αυτό. Και αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι οι περισσότεροι από του συμμετέχοντε δεν ήταν κατά της ιδέας ε, αυτής καθεαυτής της μεταφοράς δικαιωμάτων, αλλά ε, θεώρησαν ότι το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αποφασίσει πώς και πότε θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση, την οποία θα πρέπει εδώ να σας διαβάσω. Κυρία Πρόεδρε, και εσείς η ίδια αναφερθήκατε Το γεγονός ότι ε, πλέον ε, έχει ξεκινήσει η ισχύ της Συνθήκη της Λισαβόνας, ε, υπάρχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις για κάθε θεσμικό όργανο και φυσικά υπάρχει και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας. Όπως σας έχω ήδη πει, πράγματι η συνθήκη της Λισαβόνας θα έχει πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες ε, στην ε, πλήρη εφαρμογή της και θα πρέπει να σεβαστούμε τα όσα γράφονται στους κανόνες ε, της συνθήκης. Ξέρω ότι ετέθησαν κάποια θέματα στους προκατόχους μου στην Ισπανική και στη Σουηδική Προεδρία και θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σεβαστή η συνθήκη όχι μόνο στο γράμμα της αλλά και στο πνεύμα της. Δεύτερον, όντως μπορούμε ε, να συνεργαστούμε με επικοδομητικό τρόπο. Το προσωπικό μου και οι υπόλοιποι μπορούν ε, να σας διαβιβάζουν πληροφορίες και θα φροντίσουμε να είστε πάντα καλά ενημερωμένοι. Γνωρίζω την άποψή σας για το θέμα των διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή σας ως παρατηρητές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσδώσει κάποια σαφήνεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε όλοι από κοινού επικοδομητικά. Ε, κοιτάζω εδώ αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις ε, οι οποίες μετέθησαν. Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι κάλυψα τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία ετέθησαν και θα ήθελα τώρα να ακούσω τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη του Κοινοβουλίου που έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν είναι πολλοί. Ελπίζω να σεβαστούμε την ώρα στις 10 και 4. Κύριε Στίβενσον, κύριε Μπιλμπάου. Καταρχήν... Και σαν σας προσέδω. Ο κύριος Στίβενσον καταρχήν, ο αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που έχετε αυτή την καθήκη θέση για την μεκροκρομπική κατάσταση. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κάλεκερ, όμως αυτά τα μακροπρόθεσμα θέματα ε, δεν αποτελούν τμήμα των συνθήκων προσχώρησης της Ισλανδίας, ενώ εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα, καθώς οι ε, Ισλανδοί είναι ε, η κυρία επιχειρηματική δραστηριότητα που θα επιφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν καταστούν μέλη. Δεν ε, θα πρέπει να επιτρέψουμε να λειτουργούν με ανευθυνό τρόπο, γιατί δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στο πώ θα του καλωσορίσουμε εμεί ω πλήρη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τάκια τη ποσοστώσης. Άκουσα τι είπατε για τη συνεργασία μεταξύ ελαιών και επιστημόνων. Εγώ ε, είδα ότι το ISIS ε, ε, φέτος το χειμώνα, μάλλον συγγνώμη για τις συζητήσει ε, του χειμώνα, εξέδωσε κάποιες προκαταρκτικές συμβουλές, όμως είδαμε ότι η θνησιμότητα ε, των ψηριών αυξήθηκε ενώ η αναπαραγωγική βιομάζα παρέμεινε σταθερή και συνιστά το ΆΙΣΕ σε περαιτέρω περικοπές ε, στα προηγούμενα έτη. Είχαμε μείωση των αριθμών των ημερών ε, αλία στη θάλασσα και παρόλα αυτά είδαμε να αυξάνεται η θνησιμότητα. Έτσι λοιπόν το να έχουμε περικοπή των ημερών στη θάλασσα δεν έχει αποτέλεσμα. Ξέρω ότι η μεταρρύθμιση ε, να ζητά την εξέβρεση εναλλακτικών συστημάτων, όμως ε, από ό,τι φαίνεται η περικοπή στην ελευτική προσπάθεια, στην ελευτική δραστηριότητα φέτος το χειμώνα δεν πρόκειται να έχει ουσιαστικά αντίκτυπο στην εθνισμότητα των ψαριών. Πρέπει λοιπόν να ξεύρουμε άλλες προσεγγίσεις επιπρόσθετα. Ε, δεν ε, ε, επαρκούσαν τα όσα είπαν οι επιστήμονες και το και το ISIS αυτό. Είπε ότι δεν μπορούν να δώσουν μια κατάλληλη ανάλυση των αποθεμάτων για τρεις κρατη κράτη-μέλη και ειδική σας χώρα και η Γαλλία και οι κάτω χώρες δεν έχουν ε, ουσιαστικά αποκαλύψει ε, ένα κατά προσέγγιση νούμερο για τις απορρίψεις. Έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατό να γίνει η επιστημονική ανάλυση. Και τώρα λοιπόν σας παρακαλώ να δυσφαλίσετε ότι και η δική σας χώρα αλλά και οι Γαλλία και οι 100 χώρες θα παράσχουν αυτές τις πληροφορίες για τις απορρίψεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλύτερα συμπεράσματα πριν να επιβάλλουμε περαιτέρω περικοπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, ε, να σας πω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην αποδοτικότητα και στην εφορία. Όμως, αν ε, δούμε στο παρελθόν ότι αυτή η εξίσωση μπορεί να φαίνεται απλή, δεν είναι. Και δεν είναι γιατί λαμβάνοντα υπόψη τις δυνατότητες ε, που είχαμε να λύουμε το, γάδο, το γάβρο μας στο βορρά ή το μερλούκιο, είδαμε ότι η απαγόρευση αλίας ε, δεν έχει θετικά αποτελέσματα στο απόδομα. Έτσι λοιπόν πρέπει να τα έχουμε αυτά υπόψη όταν μιλάμε ε, για την αποδοτικότητα και για την αηφορία. Επίσης, εσείς μιλήσατε για συνεργασία μεταξύ επιστημονικού τομέα και λέω, εγώ πιστεύω ότι όταν παρουσιάστηκαν αυτά τα εργαλεία, αυτό ήταν δυνατό και θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στο θέμα του γάβρου, που αποτελεί ένα παράδειγμα που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον τουλάχιστον ε, στη χώρα μου και στην περιφερειά μου, ο ίδιος ο κλάδος ενδιαφέρεται περισσότερο από όλους για να έχει ε, ε δραστηριότητα, γιατί κοιτάξτε το μόνο που ξέρουν να κάνουν για να ζήσουν είναι να αλλιεύουν. Έτσι λοιπόν θα σας ζητούσα αυτή ε, η επιστημονική συνεργασία με τον κλάδο ε, να λάβει χώρα και σε θεσμικό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να εργαστούμε με μεγαλύτερη διαφάνεια και εμείς ε, εδώ από το Κοινοβουλίο με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Γιατί αν κάτι με εξέπληξε εμένα, ήταν η έλλειψη διαφάνειας με την οποία εργαζόμαστε ενίοτε όταν φτάνουν το πράγμα στο Συμβούλιο. Το λέω με απολύτη ειλικρίνεια γιατί πραγματικά αυτό έζησα και αυτό με λυπεί και αυτό αισθάνομαι. Ε, τα κράτη ε, ουσιαστικά ασκούν τέτοια εξουσία και έρχονται να ε, αλλάξουν και να τροποποιήσουν τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν επιτάπητος. εγώ έχω εργαστεί σε θέματα διαφάνειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ζητήσω και εσείς να εργαστείτε για την επιτεύξη της διαφάνειας για να έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια. Δεν μπορούμε να ζητάμε μεγαλύτερη συνεργασία από τον τομέα και να μην έχουμε εμεί την ίδια συνέπεια και την ίδια στάση σε διοργανικό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο. Τρίτον, δεν ήταν το σαφρίδι το μόνο είδος για το οποίο είχαμε συνεργασία των επιστημονικών Ινστιτούτων και του ελευτικού κλάδου. Στο θέμα του Γαύρου, επίσης, ε, υπήρξε συνολική συνεργασία μεταξύ του ελευτικού κλάδου, των επιστημονικών ιδρυμάτων και στην περίπτωση αυτή του Ισπανικού Ινστιτούτου και του Άσκη που είναι ε, ένα ίδρυμα στη χώρα των Βάσκων ε, και ε, αυτό το σχέδιο που εκπονήθηκε είναι καρπός αυτής της συνεργασίας, δηλαδή της συνεργασίας των Ιδρυμάτων με τον λευτικό κλάδο, καθώς ήθελαν να καταστήσουν αυτήν την ελευθερική δραστηριότητα αποδοτική. Επίσης, θα ήθελα να σας ζητήσω να εργαστείτε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία για να δώσετε ένα μεγαλύτερο κύρος στο ρόλο των αλλιέων. Κάθε φορά που μιλάμε για την αλληλεία, δίνουμε μια αρνητική εικόνα των ατόμων που αλλιεύουν. Ε, και εγώ νομίζω ότι στο πρόγραμμά σας θα έπρεπε να συμπεριλάβετε ε, ουσιαστικά και μια πραγματικότητα η οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Και όταν μιλάμε για έλλειψη επιστημονικών δεδομένων, δεν είναι αυτό πάντοτε πρόβλημα του κλάδου, δεν είναι πρόβλημα των αλλιέων. Έτσι λοιπόν θα συζητούσα να το πράξουμε αυτό και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, είμαι συγγήτρια για το μακροπρόθεσμο σχέδιο για το γάβρο, το μόνο που κάναμε ήταν ένας τριμερής διάλογος ε, για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και δεν θέλω να το σχολιάσω περαιτέρω. Εγώ έφτασα σε μια αρκετά προχωρημένη θέση με την Ισπανική Προεδρία, όταν μας ανακοίνωσαν ότι είχαν αμφιβολίες για την ε, νομική βάση και την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εσείς πιστεύετε μπορούμε να καλέσουμε ένα τρεμερή διάλογο το Σεπτέμβριο έτσι ώστε να δώσουμε μια οριστική όθηση σε αυτό το σχέδιο, γιατί το αναμένει τόσο ο τομέας, γιατί συνέπεια ήταν ότι φέτος για μια ακόμη φορά αντί να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο υπήρξε μια απόφαση της ε, του Συμβουλίου μετά από πρόταση της Κομισιόν και ακριβώς ε, ε, ουσιαστικά πρόθεσαν αυτό που ήθελαν να αποφύγουν με αυτό το σχέδιο. Και θα ήθελα να μας πείτε και ε, πώς θεωρείτε ότι ε, θίγεται η εμπορία ε, στον τομέα και ποιες είναι οι συνέπειες για τις ευρωπαϊκές αλευτικές ε, επιχειρήσεις γιατί υπάρχουν ε, πάρα πολλά παράπονα σε σχέση με τον έλεγχο που γίνεται με την εποπτεία στις τρίτες χώρες. Κυρία Σάντσε, ε, για να έχει χρόνο να απαντήσει ο Υπουργό, σα παρακαλώ να είστε σύντομο. Να ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την παρέμβασή του. Για... Από τις προτεραιότητες που αναφέρατε, εγώ θέλω να τονίσω τη δημοσιονομική προτεραιότητα ε, αν ε, έχει σημασία η αλία δεν πρέπει να δούμε περικοπές στον προπολογισμό, θα πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό για την αλία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τίθεται ιδιαίτερα το θέμα. να φερθεί στη συνεργασία μεταξύ ε, του αλευτικού κλάδου και των επιστημονών. Εγώ νομίζω ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την ερασιτεχνική αλία και υπάρχει και μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή ότι θα πρέπει να γίνει μια διερεύνηση στην αλυσίδα της αξίας προκειμένου ε, να ξέρουμε ποιε είναι οι δομές της αγοράς ε, και επίσης θα πρέπει να δούμε αν γίνεται σωστή διαχείριση από το αλληλευτικό ταμείο. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό δρόμο για να ενισχύσουμε και τη σχέση με τα τρίτα κράτη. Εγώ νομίζω ότι ο οδό τη ε, αηφορία, ε, αν ε, εισαγάγουμε εκεί και τι σχέσει με τι τρίτε χώρε, μπορεί να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οδό. Θα ήθελα επίση να επιστήσω την προσοχή σα στο αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον ελεκτικό τομέα, ε, καταρχήν ε, για τις εμπορικές σχέσεις ε, πρέπει εσείς να τονίσετε τη σημασία που έχει η Αλία σε αυτές τις εμπορικές σχέσεις και να έχετε κατά νου και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου να υπάρχει ισορροπία δηλαδή σε αυτό και δεύτερον νέες ελευτικές δραστηριότητες, νέες ελευτικές ευκαιρίες ε, έχουμε και την ε, πολιτική γυτνίασης και θα ήθελα να αναφερθώ και στο Μαρόκο γιατί το Φεβρουάριο θα λήξει η συμφωνία και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε τις κατάλληλες βάσεις για μια, μια συνέχιση της συμφωνίας. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στις τελευταίες ερωτήσεις και κατόπιν μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη του Κοινοβουλίου για τις πολύ καλές ερωτήσεις που έθεσαν. Ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις του κ. Στίβενσον. Ήδη είπα ότι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την προσχώρηση της Ισλανδίας είναι αρκετά σημαντικά η προσχώρηση. Ουσιαστικά δεν κρίνεται από τα λευτικά ζητήματα, αλλά φυσικά τα ελευτικά ζητήματα είναι μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή στη διαδικασία προσχώρησης ε, και νομίζω ότι είναι και πολύ σαφής η θέση της Επιτρόπου. Έτσι λοιπόν ε, θα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά ε, το, τις διαπραγματεύσεις και ιδίως ε, τα θέματα που αφορούν την αλία. Τώρα, για το σύστημα των τακτικών ποσοστώσεων. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όλα τα κρατημέλη να σέβονται τις υποχρεώσεις τους από το σημερινό σύστημα, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε ίσως κανόνες για όλους και όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι στη μελλοντική κάλπο αυτό θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα περιλαμβάνεται και ήδη σας ανέφερα τι συζητήθηκε στο Βίγκο και ποια είναι η τοποθέτηση των συναδέλφων ε, για τα τάκια και τις Εγώ άκουσα τις παρατηρήσεις σας σχετικά, αλλά Πιστεύω ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη υποστηρίζουν τη διατήρηση των τακτικών ποσοστώσεων. δηλαδή και το σημερινό καθεστώς για αυτό το συγκεκριμένο φάκελο. Τώρα να περάσω στην κυρία Μπιλμπάου. Σωστά αναφερθήκατε στο θέμα της ε, κερδοφορίας και των τιμών. Επίσης, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, δίκιο έχετε. Και εγώ είμαι θιασότης αυτής της προσέγγισης. Δεν ε, έχουμε μόνο το θέμα του σαφριδίου, φυσικά έχουμε και το θέμα του Γαύρου. Υπάρχουν προβλήματα και εκεί και αναφερθήκατε και στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι αλληλείς. Ξέρω ότι είστε ανυπόμονοι και θέλετε να σημειωθεί πρόοδο στο θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να σα ζητήσω λίγη υπομονή ακόμη. Εργαζόμαστε εντατικά επί των θεμάτων αυτών και φυσικά σημειώσαμε και τις προτάσεις σας. Έτσι λοιπόν θα επανέλθουμε αργότερα σε αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε να ξεβρούμε μια ρεαλιστική λίστα το συντομότερο. Τώρα, Κύριε αναφερθήκατε σε θέματα προπολογισμού. Εγώ δεν τα ανέφερα, αλλά φυσικά και είναι σημαντικά. Αν ε, θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη ελευτική πολιτική, χρειαζόμαστε και τους κατάλληλους πόρους. Και ξέρω ότι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, δεν προβλέπονται αυξήσεις στον προϋπολογισμό αλλά θα προσπαθήσουμε να έχουμε τους κατάλληλους πόρους διαθέσιμους έτσι ώστε να έχουμε η φοροαλία. Επίσης, πολύ σωστά αναφερθήκατε ε, στην εραστεχνική αλία, στην αλία μικρής κλίμακας ε, και θέλουμε, να θέλουμε και εμείς να δώσουμε σημασία σε αυτό το θέμα στο Συμβούλιο. Αυτή η αλία μικρής κλίμακας ε, εντάσσεται στη συζήτηση. Επίσης, ε, συζητήσαμε και τον ορισμό του small scale fishing. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα βέβαια η συζήτηση, αλλά πολύ σωστά αναφερθήκατε εσείς ε, σε αυτό τον αρέσει τεχνικό στόλο. Επίση, αναφερθήκατε και στι ε, εμπορικέ συμφωνίε με τρίτε χώρε. Και κάνατε λόγο και το Μαρόκο. Το σημερινό πρωτόκολλο λύγει στα τέλη Φεβρουαρίου του 2011. Αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντική για αρκετά κράτη-μέλη και επίσης ε, και από δημοσιονομική σκοπιά είναι σημαντική συμφωνία. Όμως, ε, όπως ξέρετε, με κάθε συμφωνία γίνεται μια μελέτη αξιολόγησης και αναμένουμε τα πορίσματα αυτή της μελέτης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και φυσικά εμείς ε, σεβόμαστε το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Κομισιόν Προεδρία και αναμένουμε να δούμε τι θεωρεί ότι είναι σκόπιμο η Κομισιόν ε, σε ό,τι αφορά την ανανέωση της συμφωνίας αυτής. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, Πρόεδρε, και σημείωσα και προτάσεις που έγιναν. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας γνωστοποίησαμε λοιπόν τις ανησυχίες της Επιτροπής Αλίας. Θα ήθελα να απαντήσω σε μια ερώτηση που θέσατε εσείς για την ε, τροποποίηση του κανονισμού 2187 για τα τεχνικά μέτρα για τη Βαλτική θάλασσα, τα οποία ε, θα πρέπει να, εθε, να τεθούν σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου για να μην υπάρχει νομικό κενό. Δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία πριν από το Δεκέμβριο. Θα καθορίσουμε ε, συντονιστή και θα συζητήσουμε το θέμα το συντομότερο δυνατόν. Επομένω, να σα διασκεδάσω τι ανησυχίε σα εδώ και να σταθώ και σε ένα θέμα το οποίο επισημάνθηκε και είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή Αλία και κανένα δεν γνωρίζει πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο έκανε τέτοιε περικοπέ στο Συμβούλιο, στον προπολογισμό Αλία ουσιαστικά μείωσε όλες τις γραμμές προϋπολογισμού και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις με πολύ ψηλά ποσοστά και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο και αδικαιολόγητο να γίνεται κάτι τέτοιο. Κανένα στον τομέα δεν θα μπορέσει να κατανοήσει για ποιο λόγο γίνονται περικοπές αυτή τη στιγμή όταν είμαστε σε πλήρη συζήτηση για την ε, μεταρρύθμιση. Ε, και είναι απαραίτητο να έχουμε επιπλέον πόρους, όχι να μας κόψουν και αυτούς που έχουμε. Και επειδή ε, στο παρελθόν ε, το ε, Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο στις μη υποχρεωτικές δαπάνες, και ενώ τώρα δεν έχουμε, θα ήθελα να σας ζητήσω να προσέξετε ιδιαίτερα στο θέμα, ώστε να αυξηθούν τουλάχιστον τα ποσά στα αρχικά κονδύλια που είχαμε. Το Κοινοβούλιο, κύριε Προεδρεύοντα, μετά από όλα αυτά σας προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του και περιμένει να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα ε, στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Διακόπτουμε για δύο λεπτά για να συνοδεύσουμε τον Υπουργό μέχρι την πόρτα τουλάχιστον. Eh, λοιπόν, είμαστε λίγοι βέβαια στην αίθουσα, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό λοιπόν να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι το θέμα το οποίο ανέφερε και ο Υπουργός και το οποίο απάντησα εγώ στο τέλος, η τροποποίηση του κανονισμού 2187-2005 για την ε, πρόληψη για τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα στη Βαλτική θάλασσα. Είναι τα τεχνικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να διαχωριστούν φέτος από την απόφαση για τα τάκτη και τις ποσοστώσεις, διότι βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να αποφασίζονται μέσω συναπόφαση και θα είναι εκτό ε, τα και ποσοστώσεων και χθε ε, στη συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίσαμε επειδή το θέμα είναι κατεπήγον και για να μην υπάρχει κανένα νομικό κενό την 1η Ιανουαρίου του 2011 θα πρέπει να εργαστούμε ταχύτατα και ε, η ομάδα του κυρίου Γκόρμπατσεφ και του κυρίου Στίβενσον πήραν αυτή την ε, έκθεση. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει την πρόταση. Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος ε, από όσους ε, είναι εδώ από την Κομισιόν. Ε, πλησιάζουμε τις διακοπές και εξαφανίστηκαν όλοι. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Θέλω να σας κάνω μία σύντομη εξήγηση. Η, ο κανονισμός για τα τάκτη τη συνδέεται με τεχνικά μέτρα. Πέρυσι είχαμε συμφωνήσει τον Οκτώβριο σε ένα μέτρο ο συνθήκης της Λισαβόνας. Εφέτος βέβαια ο κανονισμός για τα τάκ της Βαλτικής πρέπει να συνάδει με τη συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή ε, μπορούν να ε, αναφέρονται μόνο οι διατάξεις για τις αλληλευτικές δυνατότητες και προτείνουμε να υπάρξει μία τροποποίηση των ε, μέτρων για να περιληφθούν μόνο αυτές ε, οι δύο διατάξεις ή στον κανονισμό. Δηλαδή, καταρχήν, ε, μία διάταξη σχετικά από τις απορρίψεις και τις νόμιμες αφήξεις πλοίων σε σχέση με ε, τις ε, περιοχές ε, όπου αναπαράγονται τα ψάρια και αυτό θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και επίσης θα ήθελα να σας πω προς ενημέρωση ότι όλοι οι κανονισμοί για τα τεχνικά μέτρα σχετικά και με τη Βαλτική Αμερική θα αναθεωρηθούν στην επόμενη κοινή αλλιευτική πολιτική, άρα αυτό θα συμπεριλάβει και μία αναθεώρηση του κανονισμού των ΤΑΚ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει το λόγο επί του θέματος. Φαίνεται ότι όχι. Ωραία λοιπόν. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επειδή το θέμα είναι κατεπήγον και όπως είχαμε συμφωνήσει εχθές επιμένω σε αυτό ε, πρέπει να γίνει τα πάντα γρήγορα. Θα παρουσιαστεί το σχέδιο έκθεση 29 Σεπτεμβρίου, προθεσμία 20 Οκτωβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 26-27 Οκτωβρίου και θα πάει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου για να προλάβουμε ε, το χρονοδιάγραμμα που έχουμε κάνει είναι λίγο περιορισμένο το ε, χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζω να προχωρήσουν ε, γρήγορα τα πράγματα και να περάσουν τα πάντα, όλα τα στοιχεία στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της σας διάταξης, μία παρουσίαση μιας μελέτης σχετικά με την πρόληψη των παρεπιπτόντων αλλιευμάτων και των ειδών στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη αυτή είχε ζητηθεί στην προηγούμενη θητεία από τους σοσιαλιστές το αποφάσισε η Επιτροπή Αλληλείας ε, της προηγούμενης θητείας και έχει γίνει από το Irish Fishing Board ε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Σαντάντριους ε, και ο κύριος Ράιαν θα κάνει την παρουσίαση που είναι υπεύθυνος για την θαλάσσια τεχνική του Irish Fisheries Board Έχετε το λόγο, έχετε όσο χρόνο στη θέλετε στη διάθεσή σας. Εμένα μου έγραψαν 20 λεπτά, αλλά μπορείτε να μιλήσετε για όσο θέλετε, αρκεί φυσικά να μην υπερβείτε πάρα πολύ το χρόνο αυτό. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ω συνήθως τεχνικά προβλήματα. Θα σας κάνω μια παρουσίαση για μια μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε προσφάτως ε, και είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα στα κοιτοειδή. Είναι μια μελέτη που κάναμε εμείς στην Ισλανδία σε συνεργασία με, το Πανεπιστήμιο Σαντ Είμαι επικεφαλής ε, του ε, τμήματος αλληλευτικών εργαλείων στο Ινστιτούτο της Ιρλανδίας. Θα σας δώσω μια εικόνα λοιπόν του προβλήματος των των αλληλευμάτων. Αυτός ήταν ο στόχος της μελέτης που μας ζητήθηκε και θα δούμε από εκεί και πέρα κατά πόσον υπάρχει αποτελεσματικότητα από πλευρά κόστου ε, στο σύστημα το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν κάποια συμπεράσματα και ε, συστάσεις τα παρεπιπτόντα ανταλλαγματα είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Διαπιστώσαμε ότι είχαμε κάποια ε, ε, παρεμπίπτοντα και μόνο κάποιες πολύ σπάνιες ε, μεταναστευτικές ε, ε περιπτώσεις ε, για φάλαινες δεν ε, πλήττονταν από το φαινόμενο. Αλλά η έκταση και το βάθος του συστήματος ναι μένει είναι κατανοητή, αλλά δεν ξέρουμε πότε, πώς και γιατί έχουμε παρεπίπτοντα λιεύματα τέτοιου είδου. Υπάρχουν ανησυχίες για κάποια συγκεκριμένα ιδιαλίευση. Ε, πριν από κάποια χρόνια είχαμε ε, πελαγική αλληλεία. The harbor porpoise in, the Baltic Sea, where the population levels are very low level. Για κάποια είδη και είχαμε και πολλά, πολύ χαμηλά ε, επίπεδα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά πάντα εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι τα δελφίνια είναι χαρισματικά ζώα και όλοι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακριβώς λόγω της συμπάθειας που υπάρχει στα δελφίνια. Εξετάσαμε λοιπόν τον κανονισμό και τις οδηγίες που ασχολούνται με το θέμα αυτό, τον ε, ο κανονισμό 812-2004 και την οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους και προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Για την οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους, η οποία ξεκίνησε το 1998, Συγγνώμη, το 1992 υπάρχουν οδηγίες για να παρακολουθούνται τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα και να δίνονται στοιχεία κάθε 6 χρόνια. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν ε, κάλυπτε η οδηγία ε, όσα έπρεπε να καλύπτει και υπήρξε ο κανονισμός του 2004 που έχει δια, παρόμοιους στόχους. Υπάρχουν κάποιες απαιτήσει για αιτήσεις εκθέσεις εδώ και υπάρχει παρακολούθηση και ο μετριασμός των αποτελεσμάτων. Το θέμα είναι ε, κατά πόσο επετέφθησαν αυτοί οι στόχοι. Για να κατανοήσουμε το πρόβλημα, το πιο βασικό που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι σε τι κατάσταση βρίσκονται τα διάφορα είδη και στα ευρωπαϊκά ύδατα δεν είναι σαφές ε, πόσος ακριβώς είναι ο πληθυσμός και το μόνο που έχουμε είναι κάποιες εκτιμήσεις για την αυθονία τους. Ε, χρησιμοποιούνται τρεις τεχνικές, ε, ε, η συμβατική δειγματοληψία από απόσταση, μία δειγματοληψία που βασίζεται σε συγκεκριμένα μοντέλα και κάποια μοντέλα αναλύευσης. Όλα βέβαια έχουν τα υπέρ και τα κατά τους και φυσικά υπάρχουν και κάποιες διακυμάνσεις που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια των ε, μεθόδων μετρήσεων. Η ακρίβεια της μεθόδου ε, βασίζεται πάντα στο επίπεδο κάλυψης και εδώ υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Είναι σποραδικές οι καλύψεις που έχουμε και δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Έχουμε απόλυτες εκτιμήσεις για τα βασικά είδη ε, ριγχοφάλινες, μαυροδέλφινα, ζωνοδέλφινα και κάποια άλλα και έχουμε και κάποια στοιχεία για το τι έχουμε στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική Θάλασσα και στον ε, Νότιο-Ανατολικό Ατλαντικό. Αυτό βασίζεται σε τρεις ε, έρευνες, ε, τη ΚΑΝΣ 1 και 2 και μια πιο πρόσφατη η οποία αποκαλείται Κόντα. Ε, αλλά πέρα από αυτά τα βασικά είδη γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για τα υπόλοιπα είδη και για το πώς καταμερίζεται ο πληθυσμός και πώς μεταναστεύει ο πληθυσμός από τη Βόρεια Θάλασσα στον Ατλαντικό και διάφορα τέτοια στοιχεία. Και επίσης έχουμε πάρα πολύ λίγα δεδομένα για την Μεσόγειο και για τον Εύξηνο Πόντο. οι εκτιμήσεις είναι ετερογενείς και κυρίως ε, μη ικανοποιητικέ και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι όταν δεν ξέρουμε ε, πόσος είναι ο πληθυσμός με τον οποίο ε, έχουμε να κάνουμε. Να σας δώσω μία εικόνα ως προς τις κλίμακες που εξετάζουμε. Έχουμε εδώ 340.000 για όλη την περιοχή για την για το φαλιανό και κάποια στοιχεία αντίστοιχα για το άσπρο ριχοδέλφινα και για τη ριχοφάλαινα. Ε, εδώ έχουμε και κάποια στοιχεία τα οποία βλέπετε για τη ε, μελέτη της κόντα και σας δίνουν μία εικόνα για τα ποσά για τον πληθυσμό που έχουμε. Η μελέτη αυτή της IUCN είναι θεωρείται μία από τις πληρέστερες μελέτες που έχουμε για το σε τι κατάσταση βρίσκονται τα διάφορα ε, είδη. Ο Φαλιανός ε, είναι αρκετά ε, εξαπλωμένος και αυθονή στην Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική. Το κοινό δελφίνι είναι αρκετά διαδεδομένο στη Μεσόγειο. Ε, από εκεί και πέρα το ρινοδέλφινο απειλείται ε, και η ριγχοφάλαινα δεν θεωρούμε ότι βρίσκεται υπό απειλή. Ε, για όλα αυτά τα είδη, ε, σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι έχουμε επάρκεια, υπάρχουν, αυθονούν. Τώρα, για το πώ αξιολογούνται τα παρεπίπτοντα λεύματα. Υπάρχουν κάποιε μέθοδοι. Βλέπουμε τι προσαράξει, ε, συζητήσει με του αλληλεί, το ημερολόγιο σκάφου, αλλά κυρίω έχουμε άμεσε ανεξάρτητε παρατηρήσει από παρατηρητέ και ηλεκτρονική παρατήρηση προσφάτω. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστα μόνο τα άμεσα στοιχεία παρατήρησης. Ε, δεν είναι καλές προσεγγίσεις για τα παρεπίπτοντα αλεύματα ή άλλες μέθοδες. Για τα επίπεδα παρεπιπτόντων αλληλευμάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική, ε, βάσει του 8-12-2004, από τα 135 είδη κοιτοειδών που παρατηρήθηκαν, έχουμε 9.500 παρατηρήσεις είναι ασυνεπή τα στοιχεία από τον τρόπο που ε, διαβιβάζονται. Θα αναφερθώ λίγο παρα... κάτω σε αυτό. Αλλά αν τα προβάλλουμε στα επίπεδα του στόλου, έχετε τα στοιχεία εδώ που έχουμε στη διαφάνεια. Έχουμε περίπου 1.200 ε, φαλιανούς ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 500 ε, από γαλλικά δίκτυα, κοινά αδελφίνια στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και ε, κοινά αδελφίνια στην Γαλλία από πελαγικές ε, τράτες. Όλα αυτά είναι προβολές και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι σε κάποια είδη υπάρχουν προβλήματα, αλλά σε πολλά άλλα είδη που παρακολούθηκαν με, δεν είχαμε τέτοια παρεπίπτοντα αλλιεύματα σε έξι χρόνια, επομένως μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποια είδη και όχι με όλα. Τώρα, για την ε, Μεσόγειο και την έξινο πάντα, ε, πόντο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έχουμε ελάχιστα στοιχεία και πληροφορίες, έχουμε πολύ ε, λίγα προγράμματα παρατήρησης. Ορισμένες φορές δεν υπάρχει και καμία παρατήρηση και επίσης διαπιστώνονται πολύ σοβαρά προβλήματα με άλλα προστατευόμενα είδη, όπως για παράδειγμα κάποιες χελώνες. Ε, στη Μεσόγειο δεν γνωρίζουμε τίποτα για τα ε, παρεμπίπτοντα λιεύματα, αλλά υπάρχουν ενδείξεις που μας λένε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με προστατευόμενα είδη. Τώρα, για τον 8.1.12 και την παρακολούθηση και το πόσο αποτελεσματική είναι. Δεν έχουμε επαρκή δειγματοληψία, υπάρχουν προβλήματα μεταξύ ε, των κρατών μελών και τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται τα στοιχεία. Ε, υπάρχουν ε, και ενδείξεις ότι ορισμένες φορές δεν παρακολουθούνται τα κατάλληλα είδη και ορισμένες φορές είναι υπεραισιόδοξη η στόχοι παρακολούθησης και αρκετά δαπανηρή. Θα αναφερθώ και σε αυτό στη συνέχεια. Το πρόβλημα είναι ότι σε έξι χρόνια παρακολούθησης ουσιαστικά δεν έχουμε καμία αξιόπιστη αξιολόγηση για το κατά πόσον έχουμε επιπτώσει στην αυθονία των ειδών. Δεν ξέρουμε πόσα γίνονται. Υπάρχουν υποψίες ότι γίνονται κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε. Ένας από τους στόχους ε, του 812 είναι να δούμε κατά πόσον ε, επιτυχάνεται αυτός ο στόχος του 0,3. Αυτός είναι ένας αποδεκτός ε, δείκτης παρακολούθησης από στατιστικής πλευράς. Υπάρχουν και κάποιες διατάξεις στον κανονισμό που λένε ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε ένα 5 έως 10% σε πιλωτική βάση. Τα περισσότερα κάποια κράτη-μέλη καταχρώνται φυσικά αυτού του στόχου. Και βλέπουμε ότι το επίπεδο είναι ε, σε λιγότερο περίπου 1 σε 100 ε, αλληλευτικές ε, δραστηριότητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην πράξη είναι σχεδόν αδύνατον να επιτύχουμε το στόχο που θέλουμε. Ε, λέμε ότι χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση. Στις Ηνωμένε Πολιτείε χρησιμοποιούνται ε, ένα κάποια συγκεκριμένα επίπεδα τα οποία τον αποκαλούν δυνητική βιολογική αφαίρεση, εξετάζουν ένα 1,7% και εξετάζουν από εκεί και πέρα τι επίπεδο ε, παρεπιπτόντων αλλιευμάτων μπορούμε να έχουμε σε τι ποσοστό εδώ και έχουμε και κάποια επίπεδα αναφορά σε 1 με 2%. Έχουμε παραδείγματος χάρη 3.000 με 6.820 Φαλιανούς ε, που θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι είναι επίπεδο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο και αντίστοιχα ένα επίπεδο 1.400 με 3.600 κοινά δελφίνια. Εδώ έχετε μία, ένα διάγραμμα και παίρνετε ένα στοιχείο αναφοράς, ε, παίρνουμε ένα 1% επίπεδο αναφοράς χίλιων ζώων δηλαδή, και μπορείτε να είστε 90% ε, σίγουροι μετά από 100 ελευτικές δραστηριότητες ότι δεν έχουμε υπερβεί το όριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μεγάλη διαφορά στο επίπεδο παρακολούθησης για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε πρόβλημα. Θα πρέπει να φτάσουμε πάνω από το 90% μετά από τις 100 δραστηριότητες δηλαδή ε, για να έχετε ίσως μια καλύτερη εκτίμηση των περιπτώτων αλευμάτων. Αλλιώς ε, αν είστε σε χαμηλότερο επίπεδο και έχουμε μικρότερο ε, αριθμό αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Δεν ξέρετε αν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία. Ε, μιλάμε για ε, ε, μετακινούμενα ζώα και σε αλία σε διάφορες χώρες. Ποιος αποφασίζει τι θα γίνει, αν έχουμε κράτη που δεν είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βάρος απόδειξης ε, είναι στα κράτη-μέλη και αυτά θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει απειλή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δεσμευθούν ότι θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Τώρα, για το κατά πόσον θα πρέπει να μετριάσουμε τα αποτελέσματα του 8-12-2004, χρησιμοποιούμε ε, acoustic deterrent devices, που είναι μικρές συσκευές που ε, εκπέμπουν ακουστικά σήματα που απομακρύνουν κάποια είδη. Αυτές ε, οι συσκευές διατίθεται στο εμπόριο σε διάφορες παραλλαγές. Στις φωτογραφίες βλέπετε λίγο πώς είναι. Το κατά πόσον έχουν αποτελέσματα τώρα, όλα τα αποτελέσματα ε, καταδεικνύουν τα τελευταία χρόνια ότι είναι αποτελεσματικά για φαλιανούς ε, σε αλληλεία ε, με κάποια δίκτυα, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά για τα κοινά δελφίνια και για κάποια άλλα είδη δευτεριών. Άρα δεν είναι αποτελεσματικά για όλα τα είδη δελφινιών και το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά είναι κυρίως ε, πελαγική αλληλεία. Το κατά πόσον εξυπηρετούν το σκοπό τους. Έγιναν κάποιες μελέτες ε, από διάφορα κρατημέλη και εξετάζεται κατά πόσον ε, είναι ε, αξιόπιστα τα αποτελέσματα, έχουν χαμηλή διάρκεια σε κάποιες περιπτώσεις, ε, δεν γίνεται παρκής έλεγχος ποιότητας και το θέμα είναι ότι ε, φαίνεται ότι οι μπαταρίες λειτουργούν, παρόλα αυτά αυτά παρασκευάζονται από μικρές εταιρείε και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικά. Τώρα, ε, παρενέργειες, ε, παραδείγματος χάρη αποκλεισμού ενό ενός κάποιου φυσικού υποτόπου, αυτά δεν έχουν αποδειχθεί και αν βασιστούμε τι να, στο τι μπορούμε να κάνουμε για τους φαλιανού δεν υπάρχουν ενδείκτης ε, ότι αποκλείεται κάποιος φυσικός οικότοπος επειδή ακριβώς χρησιμοποιούνται αυτές οι συσκευές. Τώρα, ε, κάποιες ε, ανησυχίες ως προς την ασφάλεια και τη λειτουργία τους, ε, ναι υπάρχουν, παραδείγματος χάρη χημικές διαρροές από τις μπαταρίες, ε, ορισμένες φορές μπλέκονται στα δίχτυα και θέματα χειρισμού επί των σκαφών. Ε, τα περισσότερα από αυτά, από τη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ότι μπορούμε να τα υπερκεράσουμε, αλλά υπάρχουν κάποιε εύλογε ανησυχίε. Τώρα, κατά πόσο μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχει ο κανονισμός. Ε, φαίνεται να υπάρχει μια δυνατική λύση. Υπάρχει μια συσκευή που ανέπτυξαν από κοινού η Γερμανία και η Δανία που μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε κάποια στοιχεία επί του σκάφους για να δούμε αν ε, λειτουργούν αυτές οι συσκευές. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι γραμμένος ο κανονισμός, ε, το βάρος της απόδειξης είναι στον αλία και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι αποτελεσματικό, είτε θέλει είτε δεν θέλει να το κάνει. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνει στην πράξη, είναι πολύ ε, προηγμένες τεχνολογίες και δεν ε, ξέρουμε κατά πόσον μπορούμε να το κάνουμε. Το πώς το αντιμετωπίζει ο δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, κατά πόσον υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις για αυτές τις συσκευές. Ναι και όχι έχουμε, παραδείγματος χάρη, κάποιους ε, ε, ακουστικές ε, συσκευές που αντανακλούν και όταν πλησιάζει το ζώο και επίσης έχετε κάποια δίχτυα, στα δίχτυα που είναι πολύ πυκνά και τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν με έναν ακουστικό τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να τα ακούν τα κοιτοειδή. Ε, έχουμε δοκιμάσει σε πελαγικές ε, τράτες ε, κάποια είδη διχτυών που αποκλείουν τα ζώα εκτός. Χρησιμοποιούνται κάποια τέτοια δίχτυα με ανοίγματα έτσι ώστε να μπορούν να φεύγουν τα και είδη. Επίσης πρέπει να έχουμε και κάποιες απαγορεύσεις χρονικές και σε συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι λοιπόν έχετε κάποιες ε, περιοχές όπου δεν ε, ε, γίνεται αλία με απλά διαδίχτυα και φυσικά και κάποια εναλλακτικά εργαλεία δοκιμάζονται στη Βαλτική. Τώρα όλα αυτά λειτουργούν. Κοιτάξτε, δεν έχουμε αποδείξεις για κανένα. Ορισμένα είναι υποσχόμενα. Βλέπουμε ότι με αυτά τα ακουστικά δίκτυα, παραδείγματο χάρη, έχουν υπάρξει μειώσει ε, όμως ε, μαζί με ε, βλέπουμε ότι υπάρχει και μετριασμός, ότι μαζί με το και το ειδή υπάρχει και λιγότερη ελίευση και στα εμπορικά είδη. Έτσι λοιπόν δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρήση αυτών των δικτυών υπάρχει επίσης ε, ερώτημα για την οικονομική τους, για το οικονομικό τους κόστος. Τι μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε από την ομοτισκότητα της οδηγίας ε, για τα ενδυματήματα. Εμείς ε, έχουμε κάνει κάποιες αναλύσεις από την βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανθεώρηση της GBIC ε, μπορεί να, υπάρχουν, ε, μπορεί να υπάρχει μελλοντικό αντίκτυπος ε, στον πληθυσμό και μπορεί να υπάρχουν παρενέργειες στο καθεστώς των ειδών. Αν δείτε την έκθεση, φαίνεται να υπάρχουν αντιφάσεις και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των απειλών και των πιέσεων, πριν χάρη για τις φώκες της Βόρειας Θάλασσας για τον ίδιο πληθυσμό. Κάποια κράτη-μέλη λένε ε, ότι είναι ευνοϊκά τα αποτελέσματα, κάποια άλλα λένε ότι είναι κακά. Έτσι λοιπόν έχετε διαφορετικά κριτήρια και διαφορετικές ερμηνείες και όλα αυτά περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ ε, χαμηλή ποιότητα στοιχεία για τα παρεμπιπτόντα λιεύματα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι στην οδηγία ε, για τα ενδιαφέροντα δεν υπάρχουν σαφεί στόχοι, δεν υπάρχουν καθητήριε γραμμέ για την υποβολή εκθέσεων για τα κρατημέλη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει επικάλυψη του 812, αλλά δεν υπάρχει σύνδεσμη. Επίσης, ε, ε, προσπαθούν να διαχειριστούν τα μεταναστευτικά ζώα σε μία μικρή κλίμακα χώρου και η αποπτία για τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα αγνοήθηκε. Τα περισσότερα κράτη-μέλη θεωρήσαν ότι είναι πιο εύκολο να έχουν προστατευμένες περιοχές, όμως ε, κάτι τέτοιο δεν είναι αποτελεσματικό. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα μας είναι ότι η οδηγία ε, για τα ενδιατήματα θα πρέπει ε, να ξανασχεδιαστεί στον τομέα αυτό και ίσως ε, θα έπρεπε να προβλεφθεί η προστασία των κυκλοειδών κάπου αλλού. Ό,τι αφορά τώρα την αποτελεσματικότητα του κόστους, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια αξιολόγηση του κόστους της οδηγίας υπήρχαν ε, δύο στοιχεία όμως ε, που εξετάσαμε, το κόστος ε, των προγραμμάτων παρατηρητών και το κόστος της χρήσης αυτών των ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών και το αρχικό και το ετήσιο. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα παρατηρητών, λάβαμε από τα κράτη-μέλη πληροφορίες για 9.500 ημέρες συνολικά. Είχαμε τον αριθμό των των λευμάτων στα 135 ε, και είδαμε ότι το κόστος είναι περίπου 5.307.000 ε, ευρώ, όμως ε, δεν αντικατοπτρίζει το κόστος ένα ζώο την πραγματική αξία. Έτσι λοιπόν, ενώ φαίνονται τρομακτικά τα νούμερα, δεν μας λένε την πραγματική αλήθεια, την πλήρη αλήθεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές, ε, βλέπετε εδώ μια δεκίμωση από 6 σε 30.000, σε 13.000 με και αν δείτε το ετήσιο κόστος ε, και το κόστος ανανέωσης, Μία μελέτη έδειξε ότι μπορεί να έχουμε ε, από 484.000 πιθανότητα είναι περί τα 3.000 ευρώ ετησίως ε, το κόστος αν ε, χρησιμοποιηθούν σωστά οι συσκευές αυτές. Έτσι, λοιπόν, είναι υψηλό το κόστος των παρατηρητών και χρειάζεται εδώ καλύτερο συντονισμός. Πρέπει επίσης να διερευνήσουμε το θέμα νέων τεχνολογιών σε ό,τι αφορά το CCTV, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη, καλύτερα στοχευμένη η χρήση των παρατηρητών και σε ό,τι αφορά τα μέτρα μετριασμού, οι ίδιες συσκευέ είναι ακριβές και υπάρχει εδώ και μεγάλο κόστος ε, για την παρακολούθηση και δεν ξέρουμε ποιον βαρύνει το κόστος αυτό. Έτσι λοιπόν για να κλείσουμε. Ο 812 πετυχαίνει τους στόχους τους εν μέρει ναι, Σίγουρα έχει βελτιώσει τη γνώση σε σχέση με τα παρεπιπτόντα αλλιεύματα των κετοειδών και αν δει κανεί αυτήν την οδηγία και τι εκτιμήσει που έχουμε, βλέπουμε πού είναι τα προβλήματα και πού δεν έγκυται προβλήματα. Αλλά θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Δεν υπάρχει μετά από έξι ε, χρόνια ε, κάποια βάσιμη αξιολόγηση του αντικτύπου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αποτελεί ένα patchwork ε, ε, παρακολούθησης και δίνεται υπερβολική έμφαση στα μέτρα του μετριασμού σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα αντιαιτήματα, αν πετυχαίνει τους στόχους της, όχι στην πραγματικότητα. Και θα έπρεπε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά είναι αντιφατική και προκαλεί σύγχυση, έχει επικαλύψεις και ε, τελικά τα στοιχεία είναι φτωχά σε ποιότητα και ασυνεπή. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση για τη Μεσόγειο και τον Ευξηνοπόντο. Πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός για να συμφωνήσουμε για το καθεστώς του πληθυσμού τι αξιολογήσει χρησιμοποιούμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε επί στόχων ε, διατήρησης. Πρέπει να θεθούν κάποια όρια παρελευμάτων. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία και συντονισμό τη εποπτείας, τη παρακολούθησης. Ε, δηλαδή, ε, το να κάνουν κάποιοι άνθρωποι τέτοια πράγματα δεν ε, είναι αποτελεσματικός προς το κόστος. Επίσης ε, θα πρέπει η παρακολούθηση να μπει σε ένα ευρύτερο ε, πλαίσιο για το οικοσύστημα και τις παρακολούθηση της αλίας και χρειάζεται να έχουμε και νέες τεχνολογίες παρακολούθησης όπως σας είπα για το CCTV προηγουμένως. Πρέπει επίσης να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε ε, τις συσκευές, αν, αν μπορούμε να έχουμε συσκευές καλύτερες από τις ακουστικές αποτρεφτικές συσκευές, ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τα εργαλεία που να εξυπηρετούν το στόχο μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα υπόλοιπα προστατευμένα είδη, όπως παραδείγματο χάρη τις χελώνες, αλλά και άλλα είδη που θα πρέπει να παρακολουθούμε. Θα πρέπει να υπάρχει σαφή σύνδεση μεταξύ του 812 και τη οδηγία για τα ενδιατήματα και όπως σας είπα ε, πρέπει να ε, αφαιρέσουμε την ανάγκη της παρακολούθησης των περιπτωτών ελευμάτων υπό την ε, οδηγία για τα ενδιατήματα. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Eh. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ράιν για την παρουσίασή σας και μπορώ να πω ότι εμένα αυτό το θέμα, παρόλο που δεν με ενδιέφερε, θεώρησα ότι η δική σας παρουσίαση, οι συστάσεις σας και τα συμπεράσματά σας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα κατόπιν όλων αυτών δεν ξέρω αν κάποιος θέλει το λόγο. Κύριος Βαλέσσα. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι σύντομα θα φύγω, αλλά πριν φύγω θα ήθελα να αναφερθώ τη Βαλτική, διότι δεν βλέπω να υπάρχουν θέματα σχετικά με τις φώκες ε, ε, και ούτως ή άλλως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν μόνο δύο είδη και δεν ξέρω πώς εκεί μπορούμε να λάβουμε υπόψη ε, το παρεπίπτον αλίευμα και ε, τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Τι κάνουν δηλαδή τα κράτη-μέλη για να μειώσουν τα παρεπίποντα ε, ε, ε αλλιεύματα αυτού του είδους. Πρόκειται για ένα μικρό είδος και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται στις περιοχές όπου υπάρχουν μεγαλύτερες τέτοιες ε, ποσότητες ε, που θα έπρεπε να προστατευθούν Επειδή δεν έχουμε στοιχεία σχετικά με τη Βαλτική, ενώ έχουμε ε, σε άλλες περιπτώσεις, νομίζω ότι καλό θα ήταν να προσέξουμε αυτή την αλληλεία και όσον αφορά τον κανονισμό 112 του 04 δεν λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό κόστος που είναι πολύ υψηλό για την Πολωνία γι' αυτό και είχαμε ε, καταρτήσει ένα πρόγραμμα παρακολουθήσεως ε, και στην ε, διάρκεια αυτής της περίοδου δεν είδαμε αυτά τα θηλαστικά να ε, παρουσιάζονται εις ε, την περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανονικά πρέπει να παρουσιάσει, έπρεπε να έχει παρουσιάσει μέχρι το 2009 στο Συμβούλιο και εις την ε, και ε, στο Κοινοβούλιο τα στοιχεία σχετικά με τις ε, φώκες και τις, τα άλλα είδη τα οποία υπάρχουν, τα δελφίνια τα οποία υπάρχουν. Θα δώσω το λόγο, το λόγο στον κύριο Ράιαν για να δούμε αν θα μπορέσει να απαντήσει. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι βιολογικός ε, εμπειρογνώμονας ε, και τα προβλήματα της Βαλτικής είναι συγκεκριμένα. Πρόκειται για ένα μικρό πληθυσμό και ουσιαστικά και ε, πρόκειται ε, για καταστροφικές επιπτώσεις βέβαια αλλά ε, όσον αφορά τα δίχτυα στη Βαλκική υπάρχει ένα περίπλοκο πρόβλημα το οποίο δεν θα προσπαθήσω να επιλύσω διότι είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει χάσαμε την, στην διαφωνία που είχαμε και έτσι αυτή είναι η κατάσταση και ούτως ή άλλως η ιδέα μας στην ε, ε, Βαλτική δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Ε, όπως σας είπα δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας. Um, good morning. Um, Καλησπέρα σας καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τον κανονισμό 812, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι την πρώτη έκθεση σχετικά με τον κανονισμό αυτό βάσει ε, των αξιολογήσεων των κρατών μελών και όσον αφορά τη Βαλτική Όντως έχουμε ζητήσει μία επιστημονική αξιολόγηση από την ISIS και Μέχρι στιγμής δεν έχουμε συγκεντρώσει όλα τα αναγκαία ε, ε, στοιχεία. Αυτό δε που αποφασίστηκε ή μάλλον με συγχωρείτε ε, ξέχασα ότι πρέπει να υπάρξει και μία δεύτερη έκθεση επί του κανονισμού αυτού που καταρτίζεται αυτή τη στιγμή και θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου στην, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ε, στη συνέχεια της μελέτης του 2004 θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα και τα επόμενα βήματα και αυτό που παρουσίασε σήμερα ο Ντομινίκ ε, σήμερα είχαμε ζητήσει από το ISIS ε, να γίνει η αντίστοιχη αξιολόγηση στις εκθέσεις των κρατών μελών και ε, λαμβάνουμε υπόψη και άλλες μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Η κυρία Ρόμπουστ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, αλλά ε, αισθάνομαι ενοχλημένη διότι βλέπω ότι χρειάστηκε να πείτε πάρα πολλές φορές δεν έχουμε ενημερωμένα στοιχεία. Με ανησυχεί πολύ και σας ρωτώ διότι πολλές φορές ακούω όταν μιλώ με επιστήμονες ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας κατά τρόπον ώστε να να υπάρξει μια καλύτερη βάση δεδομένων. Ο κύριος Στίβενσον. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, αλλά μας είπατε ότι όσον αφορά τα κοιτοειδή ε, παραεπίπτοντα λιεύματα ε, είναι χαμηλά, αντιλαμβάνουμε ότι είναι πολύ σημαντικά και συζητούσαμε για τον ειρηνικό με την αντιπροσωπεία αυτής της Επιτροπής και ιδίω όσον αφορά τα δελφίνια κατά την αλία του τόνου ε, στην περιοχή εκείνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσπάθεια προσπαθούν ε, να απομακρύνουν από τα δίχτυα τα δελφίνια και πολλές φορές ε, και οι βουτυχτές που ε, ενεργούν σε αυτά τα πλαίσια σκοτώνονται. Δηλαδή κάνουν πολλές προσπάθειες ενώ εμείς εδώ κατακρεουργούμε πολλά κοιτοειδή. Μου φαίνεται ότι είναι κάτι το απαράδεκτο. Ελπίζω ότι σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί ε, θα λάβουμε μέτρα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, διότι εγώ ζω στην ε, δυτική ακτή της Σκοτίας, κοντά στο Φάιν και ε, όταν ήμουν παιδί βλέπαμε και φθάνανε πολλά δελφίνια που έφταναν ακολουθώντας ορισμένα ψάρια, αλλά τώρα δεν υπάρχει κανένα ε, η περιοχή έχει καταστραφεί, δεν υπάρχει κανένα ούτε ψάρι ούτε κοιτοειδές. Ε, όλα εξαφανίστηκαν και δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η κυρία Λοβέν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας, η οποία ήταν ε, πολύ πλήρης, πολύ γρήγορη βέβαια, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει πολύ αναλυτική εργασία και θα διαβάσω με προσοχή την μελέτη. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Στίβενσον, ότι κατά τη διάρκεια μου όσον αφορά όλα τα ε, κοιτοειδή ε, και τα είδη δελφινιών έχουν εξαφανιστεί, οπότε είναι ένα είδος το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε και ελπίζουμε ότι η μελέτη σας είναι ένα πρώτο βήμα προς σωστή κατεύθυνση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ την κυρία Λόβιν. Θέλετε να κάνετε κάποιο πρόσθετο σχόλιο, παρακαλώ. Σας δίνω το λόγο. Λοιπόν, έχω να κάνω διάφορα σχόλια. Ξέρω ότι οι αριθμοί είναι δυσάρεστοι, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ αναφερόμαστε σε πολλές περιοχές αλίες και σε άλλες οποίες έχουν παραβλέψει τελείως παρακολουθούμε αλληλεία από τις οποίες παρακολουθούμε για άλλους λόγους και όχι για αυτό. Πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε τα προβλήματα και πιστεύουμε ότι ε, έχουμε μια καλύτερη εικόνα τώρα για το πού βρίσκονται τα προβλήματα και πού πρέπει να δράσουμε. Έχουμε τονίσει υπερβολικά ε, λέγοντας ότι υπάρχουν ε, λύσεις, αλλά υπάρχουν λύσεις που αντιμετωπίζουν ένα είδος και ε, μία περιοχή αλληλείας. Όσον αφορά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πολλά, όντως δεν γνωρίζουμε, και τουλάχιστον ξέρουμε από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, ε, διότι Ίσως ε, οι Αμερικάνοι έχουν ε, καλά στοιχεία για την αλληλεία τους, αλλά εδώ στην Ευρώπη έχουμε αντίστοιχα, διότι από ό,τι ξέρω μπορούμε ε, να κάνουμε καλές υποθέσεις και να εστιαστούμε εκεί που πρέπει και γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτόν τον κανονισμό, ο οποίος είναι πολύ ευρύς και να παραβλέπει το ουσιαστικό θέμα. Ε, ε, Γενικώ είμαι απεσιόδοξο, αλλά ε, είμαι ακόμη πιο πολύ όταν κοιτώ τη, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλο που τώρα υπάρχει ένα, το, μια τυποποιημένη μορφή παρουσιάσεως και μπορούμε να δούμε τα στοιχεία και να διευκολύνουμε τη δουλειά μας και να γίνουν διάφορες αναλύσεις σε διάφορα θέματα. Άρα αυτό το χαιρετίζω, είμαι θετικός και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ράιν. Ευχαριστούμε πολύ και την Κομισιόν. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό το σημείο στην ημερησία διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι τα διάφορα. Υπάρχει κάτι εδώ. Ας περάσουμε τότε στο τελευταίο σημείο. Ανακοινώσεις των ε, συντονιστών έχουν διανεμηθεί αυτά. Το πιο σημαντικό είναι που θα ξαναδούμε μετά την επιστροφή μας τον Αύγουστο και θα έχουμε όλοι καιρό να σκεφτούμε επί των ε, προβλημάτων εφαρμογής συνθήκης της Λισαβόνας θα έπρεπε να έχουμε μία συνάντηση συντονιστών και των αντιπροέδρων ε, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές για να δούμε το θέμα αυτό, έτσι ώστε ο καθένας ε, να υποβάλει συγκεκριμένε προτάσεις. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται αυτά. Το μόνο που θέλω είναι να σας ευχαριστήσω. Συγγνώμη, κύριος Γκάλαχερ και μετά κυρία Ροβούστ. Κύριε Γκάλαχερ, δύο σημεία πρόεδρε. Η επόμενη συνάντηση είναι στις 30 Αυγούστου και θα εργαστούμε επί του προπολογισμού εκείνη την ημέρα. Προσπαθώ να βρω κάποιον να με αντικαταστήσει γιατί θα είμαι σε αποστολή. Πότε και τι ώρα προτείνεται να ε, συνεδριάσουμε και να ψηφίσουμε, γιατί στις 3 ίσως θα δυσκολεύονται κάποιοι να είναι εδώ και θα ήθελα επίσης να παρευρεθώ στη συνάντηση των συντονιστών σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και το Σαφρίδι, αλλά δεν θα είμαι εκείνη την ημέρα εδώ σίγουρα, γιατί έχω και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε και μία ημερομηνία το Σεπτέμβριο. Ελπίζω ότι ναι, αλλά τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες γιατί δεν τις έχω θα πρέπει να περιμένουμε να επιστρέψουμε από τις καλοκαιρινές διακοπές για να δούμε ποιες θα είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε λάβει για την ψηφοφορία στις 3. Κοιτάξτε, θα πρέπει να συζητήσω και με την γραμματεία, αλλά σας υπόσχομαι ότι δεν θα γίνει την πρώτη ώρα και ότι θα καθορίσουμε στην ημερησία διάταξη την ακριβή ώρα από τις... Ε, θα μπορούσαμε να πούμε, παραδείγματος χάρη, στις 5 να το καθορίσουμε για να έχουν ε, χρόνο οι βουλευτές να έρθουν. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι προβληματικό να έχουμε ψηφοφορία στις 3 το απόγευμα. Εντάξει, σας υπόσχομαι ότι κατά τις 5 δεν θα γίνει και την πρώτη ώρα που θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. Κυρία Ρόντουστ. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο ουσιαστικό μας πρόβλημα όσον αφορά την θέση παρατηρητού. Θα ήθελα να σας πω ότι τώρα μετά τις ε, διακοπές θα πρέπει το θέμα αυτό να τεθεί ε, εκτάκτος στους συντονιστές για να συζητηθεί και ήδη στον προγραμματισμό θα πρότεινα για την μεθεπόμενη συνεδρίαση ε, να ενσωματώσουμε το σημείο αυτό διότι αν θέλουμε να διατυπώσουμε προτάσεις θα πρέπει ε, να ε, συνδεθούμε και πάλι με τις πολιτικές μας ομάδες διότι εάν θέλουμε να αντιδράσουμε στα θέματα τα οποία συζητήσαμε χθε και δεν θέλω να επαναλάβω δημοσίως χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτικής ομάδος πρέπει να μπορέσουμε να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτό να περιληφθεί στον προγραμματισμό γιατί ε, πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στη Βρυξέλλες στις 30 Αυγούστου. Έτσι λοιπόν το μόνο που μου μένει είναι να σας ευχηθώ καλές διακοπές και τους εξαιρετικούς κύριου βουλευτέ και τους εκπροσώπους τη Κομισιόν και ελπίζω να περάσετε καλό καλοκαίρι, να φάτε πολύ ψάρι και να ξεκουραστείτε για να επανέλθετε με πολλή ενέργεια στα τέλη Αυγούστου. Τέλος της συνεδρίασης.